Okay, dear to the second half of Λοιπόν, προχωρούμε. Το δεύτερο μισό της σημερινής συνεδρίασης, σημείο 9. Είναι οι διαπραγματεύσεις ε, του ΠΟΕ για μια πολυμερή συμφωνία ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι προφανές νομίζω ότι η ψηφιοποίηση προχωρεί και αλλάζουν πολλά πράγματα και για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε τους διεθνείς κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον εντοπισμό δεδομένων, τη ροή δεδομένων, προσωπικά δεδομένα και προστασία δεδομένων και γι' αυτό ήταν πολύ σοφό από τα πολλά μέλη του ΠΟΕ, του ΠΟΕ να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ελπίζω ότι θα είναι μια επίσημη διαπραγμάτευση. Ο πρώτος γύρος έγινε 24 με 27 Σεπτεμβρίου στη Γενέβη και ο κύριος Κριστόφ Κίνερ είναι ο κύριος διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μας ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Το λέω αυτό προκατακτικά γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ σημαντικό θέμα στην εμπορική πολιτική. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος λοιπόν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργήσει μια επιτροπή παρακολούθησης που θα ασχολείται ειδικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί θα δείτε ειδικότερα ε, στην ε, παρουσίασή μου ότι ίσως καθυστερήσαμε πολύ ε, ε, ε, είναι λίγο μεγάλη το απόγευμα, αλλά θα προχωρήσω γρήγορα. Σε στενή συνεργασία με τον κύριο Ντάντι θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο μαζί σας στις σημαντικές προκλήσεις που συνεπάγεται αυτή η πρωτοβουλία. Τώρα, δύο λόγια για το ιστορικό και τη σημασία του παγκοσμίου ηλεκτρονικού εμπορίου. Μιλάμε για ε, τεράστια στοιχεία, ε, 29 τρισεκατομμύρια, πάνω από ένα δις άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για τα ψώνια τους. Ε, αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο της ε, ατζέντα, γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακά, όπου αγοράζονται προϊόντα κάνοντας κλικ στον υπολογιστή, Έχουμε και το πραγματικά ψηφιοποιημένο κομμάτι με ηλεκτρονικά προγράμματα που ανταλλάσσονται ε, διασυνοριακά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι λοιπόν πολύ ευρύτερο. Τώρα, το σημείο αφετηρίας δεν έχουμε παγκόσμιους κανόνες τώρα. Έχουμε αρχίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συντάσσουμε μια μεγάλη ατζέντα για τις ψηφιακέ διαπραγματεύσεις, αλλά δεν υπάρχουν παγκόσμιοι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό οι διαπραγματεύσει στον ΠΟΕ είναι σημαντικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολούθησε στενά το δικό μας προβληματισμό για να έχουμε μια στρατηγική. Στο τέλος καταλήξαμε με έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας πριν από δύο χρόνια που ήταν πηγή έμπνευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στην αντιμετώπιση του ψηφιακού εμπορίου. Τώρα, στον ΠΟΕ το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι ε, καινούριο θέμα και πολλοί στον ΠΟΕ τον αποκολούν νέο θέμα. Από το 1998 αρχίσαμε συζητήσεις μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για το προγραμματισμό πολυμερή επί 20 χρόνια δεν κάναμε μεγάλη πρόοδο γιατί κάποιες ε, χώρες πολύ έντονα ε, εμπόδισαν τις διαπραγματεύσεις ε, εκτός και αν θα είχαν λυθεί όλα τα θέματα της διακήρυξης της Ντόχα, κυρίως δε, θέματα που αφορούν τη Γεωργία. Μία ομάδα 17 χωρών Αποφάσισε όμως να προχωρήσει ε, με, σε πολυμερή βάση. Και η τελευταία Υπουργική Σύνοδος του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες έγινε αυτό. Μετά ακολούθησε ένας ε, χρόνος διερευνητικών συζητήσεων και μετά στο Ντάβο στην Υπουργική Σύνοδο του Ιανουαρίου φέτος μια ομάδα 17 χωρών αποφάσισαν να αρχίσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις ε, για το ψηφιακό ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως το ονομάζουν στον ΠΟΕ. Είναι ανοιχτή η διαδικασία, πολυμερής μεν, αλλά καλούμε μόνο μέλη του ΠΟΕ και περίπου 80 ε, μέλη του ΠΟΕ συμμετέχουν ε, και η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη και πρέπει να πω ότι η δουλειά είναι, που γίνεται είναι πολύ καλή. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή έχει μεγάλη οικονομική σημασία ο κλάδος, έδωσα κάποια στοιχεία, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, αυτό από πολιτικής και στρατηγικής άποψης ίσως είναι πιο σημαντικό το θέμα τώρα από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Είναι σημαντικό όχι με αυτή η πρωτοβουλία για να δείξουμε ότι η διαπραγματευτική λειτουργία του ΠΟΕ εξακολουθεί να υφίσταται και μπορεί να είναι αποτελεσματική. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό εν ώψη προσπαθειών από κάποιους να ε, ταχθούν κατά της ε, του ΠΟΕ ως φορέα διεθνούς σε σχέση με άλλους πυλώνες. Και εδώ έχω υπόψη μου την, ε, το κομμάτι επίλυσης διαφορών. Έχουμε, θα έχουμε να συζητήσουμε για αρκετές προκλήσεις στις πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Υπάρχει αυτή η τάση, θέλετε, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα χωρών και από την άλλη το επίπεδο της φιλοδοξίας παραμένει υψηλό και θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια αρχιτεκτονική αρκετά ευέλικτη που θα λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες των κρατών μελών του ΠΟΕ και βεβαίως ε, όλα αυτά πάνω στην βάση ε, του πολέμου μεταξύ ΙΠΑ, εμπορικού πολέμου μεταξύ ΙΠΑ και Κίνα που μπορεί να παρεμποδίσει τις εξελίξεις. Τώρα, για να σας δείξω τη συνθετότητα αυτών των διαπραγματεύσεων με την ε, σύγχρονη διαπραγματευτική εντολή που εγκρίθηκε στην αρχή του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε συνεκτικές προτάσεις σε κείμενο που καλύπτουν ε, αριθμό θεμάτων. Κάποια ε, εντοπίζονται εδώ, μορατόριο στους δασμούς στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις, μέτρα για την για τις συναλλαγές, εντοπισμός, ε, ο κώδικας της πηγής, ε, ουδετερότητα, ε, διατάξεις για τα spam και άλλες τα αυτόκλητα μηνύματα. Έχουμε πρόθεση να μιλήσουμε για την ροή δεδομένων και, την, και τον εντοπισμό η υποχρεωτική δημοσίευση του κώδικα πηγής, αυτό ε, οπωσδήποτε θα θέλει το Κοινοβούλιο να το συζητήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε προτάσεις ε, επίσης για την ουδετερότητα του δικτύου, επίσης ε, η, ο τομέας τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικός και έτσι πιέζομαι υπέρ ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων και πρόσβαση στην αγορά εδώ. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις επιτάπητος προφανώς, γιατί τώρα 22 προτάσεις έχουν επισήμως υποβληθεί και η Κίνα υπέβαλε μία την προηγούμενη εβδομάδα ε, θα είναι μια νέα πρόκληση αυτή γιατί κάποια στοιχεία της πρότασης ε, είναι υπερβολικά. Τώρα, για να σας δώσω μια ιδέα του πού βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτή τώρα. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Μάιο, εμείς είχαμε υποβάλει τις προτάσεις μας τον Απρίλιο. Έγιναν τρεις γύροι διαπραγματεύσεων Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και την περασμένη εβδομάδα είχαμε τον τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων όπου αρχίσαμε δεύτερη ανάγνωση των 22 προτάσεων που είναι στο τραπέζι. Η Αυστραλία ε, έκανε μια ε, έναν εξορθολογισμό όλων των προτάσεων σε ένα έγγραφο για να βοηθήσει τη συζήτηση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μια συζήτηση, πολύ θετική εξέλιξη σε σχέση με το πώς είμαστε την Άνοιξη ε, όπου είχαμε τους συνήθεις υπόπτους της χώρες του ΟΣΑ και τις προηγμένες χώρες που έχουν μεγάλη εμπειρία στο ψηφιακό εμπόριο και που συμμετείχαν. Την περασμένη εβδομάδα όμως αρχίσαμε να βλέπουμε μεγαλύτερη εμπλοκή από αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό είναι κάτι ευπρόσδεκτο, κάτι που το ενθαρρύνουμε. Είχαμε α, αφρικανικές χώρες να συμμετέχουν, η Κένια που είναι η τελευταία η Σενεγάλη, που επισήμως δεν είναι μέρος της διαδικασίας, έπαιξε πολύ δραστήριο ρόλο στις συζητήσεις. Πολύ θετικό αυτό. Είναι αλήθεια ότι την περασμένη εβδομάδα εστιάσαμε σε θέματα που είναι σχετικά τεχνικής φύσεως και όχι αμφιλεγόμενα, όπως βλέπετε και εδώ, τις ηλεκτρονικές, ε, τα ηλεκτρονικά συμβόλαια, τις υπογραφές, τις τυπολογήσεις. Όμως ε, ε, υπάρχει κάτι πολύ ευαίσθητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπερβάλλω, μια πρόταση από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία να υπάρχουν διατάξεις στο, στη μελλοντική συμφωνία για, το, για την μη διάκριση του λεγόμενου ψηφιακού προϊόντος. Αυτό είναι κάτι που συνιστά πιθανή απειλή στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπερασπίζεται και προωθεί και την πολυμορφία. Όπως ξέρετε έχουμε ένα σύστημα ποιοτικών ορίων, έχουμε ποσοστώσεις για τα καλλιτεχνικά έργα, ε, online πλατφόρμες που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις ε, ταινίες κινηματογράφου και στη μουσική και το, η αρχή της μη διάκρισης ηλεκτρονικών διαβιβάσεων ψηφιακών προϊόντων όπως τα ονομάζουν, αυτό αντιτίθεται με τοπικά στο δικό μας σύστημα της προώθησης της καλλιτεχνικής πολυμορφίας. Οπότε εδώ είμαστε σαφώς κατά και το είπαμε ηχηρά την περασμένη εβδομάδα. Η συζήτηση ήταν καλή γιατί πάνω σε αυτό το θέμα κάποιες χώρες είχαν συμφωνήσει με τις προτάσεις ε, σε άλλες περιφερειακές διαπραγματεύσεις ενώ και τώρα πέρασαν στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ενθαρρυντικό. Έκανε μια διαφορά στην διαπραγματευτική μας τακτική. Ενώ σε εύκολα θέματα όπως η διευκόλυνση ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ. Ε, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι ε, αυτά τα θέματα ε, προωθήθηκαν και δεν ήταν πολλοί εκείνοι που ετάσσονται υπέρ της ε, μη διάκρισης. Ε, αρχίσαμε να συζητάμε και για την διαφάνεια. αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δείτε σύντομα, και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια και τελειώνω με αυτό, τα θέματα για τους επόμενους δύο διαπραγματευτικούς γύρους. Πολύ εντατική είναι όπως βλέπετε. Εγώ μόλις γύρισα από τη Γενέβη την περασμένη εβδομάδα και σε τρεις εβδομάδες θα ξαναπάω πάλι για μια-δύο εβδομάδες και στο τέλος Νοεμβρίου ξανά πάλι. Τέλος Οκτωβρίου θα συζητήσω με θέματα που αφορούν ε, ροές δεδομένων, ιδιωτικότητα, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ε, θέματα που αφορούν τους πελάτες και στο τρίτη συνάντηση του τριμήνου θα μιλήσουμε για το μορατόριο στους δασμούς, ουδετερότητα δικτύου και πρόσβαση της αγοράς. Αυτά πολύ γρήγορα ε, για να σας κατατοπίσω και με χαρά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι μια μεγάλη ιστορία και μερικές φορές, κάποια φορά θα έχουμε και επιτυχία στις διαπραγματεύσεις αυτές. Είναι όμως ε, πολλά υποσχόμενα αυτά που μας λέτε ε, στην γεφύρωση του κενού ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες χώρες. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κάντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Κένερ που μας έδωσε αυτή τη λεπτομερή παρουσίαση της πρόοδου των διαπραγματεύσεων αυτών. Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες και τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες υπό το φως των νέων οικονομικών αλλαγών και των νέων τεχνολογιών. Όλοι οι σημερινοί κανόνες του πολυμερούς διεθνούς εμπορίου ε, έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τότε που δεν υπήρχε ακόμα η ψηφιακή εποχή, ήταν μόνο στην αρχή της. Άρα χρειαζόμαστε ή μάλλον έχουμε και μια μεγάλη ευκαιρία ε, λόγω των βαθιών αλλαγών που έγιναν στις ε, αλυσίδες του εφοδιασμού και στις νέες τεχνολογίες, ε, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία το, εμπορικό, ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο να γίνει μια νέα κινητήρια δύναμη των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Πρέπει να έχουμε κανόνες όσο γίνεται πιο επικαιροποιημένους και προηγμένους. Στον τομέα αυτό εργαστήκαμε επί πολλά χρόνια, ιδίω για την στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά, για να γίνει πιο αποτελεσματικό το νομικό πλαίσιο και για να δώσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα σε όλους τους εμπορευόμενους, καθώς και για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πρέπει όμως να ε, υπάρξει συμφωνία ε, ενός μεγάλου αριθμού χωρών ε, από όλο τον κόσμο ε, για τους νέους αυτούς κανόνες, ιδίως των μεγάλων ε, εμπορικών χωρών. Ε, θα πρέπει να γίνει αυτό για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια για τους καταναλωτές μας και να έχουμε καλές σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο εξορισμού είναι παγκόσμιο Άρα, αν δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες, οι κανόνες εξορισμού καθορίζονται από τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν κανόνες, πρότυπα, ε, όλο και πιο πολύ διαδομένα στην ε, ψηφιακή οικονομία. Ε, έτσι λοιπόν ε, αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για να αυξηθούν και οι εμπορικέ ροές από την Ευρώπη προς τις τρίτες χώρες. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, ε, ιδίως σε κάποιους τομείς και ιδίως για τις start-up τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη για να αναπτύξουν, να παράγουν και να ε, θέσουν στο εμπόριο προϊόντα και υπηρεσίες που θα φτάσουν σε πελάτες τους σε ολόκληρο τον κόσμο ε, και παραδείγματο χάρη στην ε, Ασία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να καταργήσουμε διάφορα μέτρα ε, που αποτελούν εμπόδιο αυτή τη στιγμή ε, για την πρόσβαση της Ευρώπης προς τρίτες χώρες. Αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να συμβάλλει ώστε να γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς οι εισαγωγές, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία μεταξύ των τελικών Ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά επίσης και σε πολλούς ε, εμπορευόμενους σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των εισαγωγών από τρίτες χώρες που γίνονται μέσω ε, ηλεκτρονικών μέσων, online. Η ασφάλεια λοιπόν των προϊόντων αυτών και η ποιότητα δεν ε, αντιστοιχούν ε, μερικές φορές ε, στα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί. Υπάρχει δυσκολία για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και άλλα διάφορα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα και που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν ασχολούνται ή εμπορεύονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, απαλύνουμε, να καταργήσουμε αυτές τις αβεβαιότητες. Τέλος, ε, στα πλαίσια του ψηφιακού εμπορίου, ε, ένα σημαντικό στοιχείο αφορά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ένα ε, asset πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι στη βάση βασικών ε, τεχνολογιών όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων, αλλά είναι και ένα πολύ σημαντικό input για διάφορες επιγραμμικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογισμικού. Γι' αυτό η ικανότητα ε, αξιοποίηση των δεδομένων για ανάπτυξη νέων πρωτοβουλειών, νέων υπηρεσιών και προϊόντων είναι ένας παράγοντας που η σημασία του θα συνεχίζει να αυξάνεται συνεχώς. Υπό την οπτική αυτή θα πρέπει να ε, εγγυηθούμε ε, στα πλαίσια να διηγηθούμε ένα διεθνές ψηφιακό περιβάλλον σαν ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί τι ίσε συνθήκε ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δημιουργούν δεδομένα, που πολύ συχνά είναι ευρωπαϊκές εταιρείε και τους ενδιάμεσου, που είναι, ε, είναι 23 χώρες και πολύ ε, πιο συχνά ε, στις ΗΠΑ, που συλλέγουν αυτά τα δεδομένα και τα αρχαιοποιούν. Αυτό είναι ένα θέμα ε, το οποίο αξίζει την προσοχή μα και αξίζει να μαθαίνουμε. Τέλος, όσον αφορά τη συμβατότητα των ε, εν λόγω ε, κανόνων με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα ε, και την ασφάλειά τους, θα πρέπει να εντοπίσουμε τον κίνδυνο μείωση των προτύπων που έχουμε φτάσει στην Ευρώπη όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια του δικτύου κλπ. Όλα αυτά τα θέματα αναφέρονται πολύ ε, σαφώς μέσα στην διαπραγματευτική εντολή και η εντολή αναφέρεται ε, σαφώς στην ανάγκη να μην τεθεί σε κίνδυνο το ισχύον ε, ευρωπαϊκό καθεστώς όσον αφορά το cyber security. Και έχουμε για το θέμα αυτό, θυμίζω, δύο πολύ σημαντικές οδηγίες από την προηγούμενη θητεία που είναι πολύ σημαντικά σημεία αναφοράς. Αυτά τα σημεία λοιπόν θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και το ίδιο ισχύει και για την ε, διανοητική ιδιοκτησία και για τα τηλεοπτικά μέσα. Ε, όλα αυτά τα θέματα, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα είναι αντικείμενο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων και γι' αυτό πιστεύω ότι η συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και το Monitoring Group θα είναι επικοδομητική και θα βοηθήσει να ε, επικρατήσουν οι δικέ μας αρχές στα πλαίσια αυτά του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπόριου. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ, κύριε για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ψυχιακή τεχνολογία έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο με πολλαπλού τρόπου μα οδηγεί σε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίε και σε νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Και τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και όλος ο κλάδο. και αλλάζει και τι ζωέ των ανθρώπων. Επομένω, είναι πολλά υποσχόμενο το γεγονός ότι οδεύουν καλά αυτές οι διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινού κανόνες στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις για την Επιτροπή. Καταρχήν, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος που παρουσιάστηκε, θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις μέχρι την επόμενη υπουργική διάσκεψη στο Καζακστάν. Ή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πέρα από αυτό που μας παρουσιάσετε σήμερα. Θα ήθελα για κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες ε, σε ό,τι αφορά τις ροές δεδομένων και την ιδιωτικότητα των δεδομένων, καθώς θα συζητηθεί τον Οκτώβριο. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά τους διευθυντές Και τέλος, ακούσαμε ότι η Κίνα παρουσίασε μια πρόταση κειμένου. Υπάρχει ήδη αξιολόγηση από την Κομισιόν για αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το Ρηνιού. Η κυρία Βερντέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την παρουσίαση Αναφερθήκατε στην ανάγκη ενίσχυση των διεθνών κανόνων σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ρυθμίσεις του τομέα αυτού. Όλοι είμαστε πεπισμένοι. Είναι ουσιαστικό για να εγγυθούμε την προστασία των δεδομένων, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση, να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι ευρωπαϊκές και να προσφέρουμε πλεονεκτήματα στου καταναλωτέ. Θέλω διευκρινήσει σε διάφορα σημεία, καταρχήν για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πώς ε, ε, νοείται να πράξετε έτσι ώστε να είναι πραγματικά ηγέτη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ευκαιρία για αυτέ. Πώ προσεγγίσατε αυτό το θέμα συγκεκριμένα για αυτέ και τι προκύπτει από τι διαπραγματεύσει, και τέλος, ο συνάδελφο, αναφέρθηκε στο θέμα της κίνα. και εγώ θα ήθελα να σας ακούσω. Ε, το κράτο αυτό έχει διαφορετικό όραμα και πρακτικές ε, σε ό,τι αφορά την τοπικότητα των δεδομένων. Ε, εδώ πώ σκοπεύετε να βρείτε μία βάση συμφωνίας. Επίσης, χαίρομαι για τη δημιουργία της ομάδας παρακολούθησης για το e-commerce. Νομίζω ότι θα είναι πραγματική ευκαιρία να εργαστούμε ευρύτερα για την ε, διεύρυνση του πολυμερούς πλαισίου και να έχουμε μια πραγματικά ενισχυμένη ψηφιακή στρατηγική. Γιατί κατά την ακρόαση του κυρίου Χόγκαν είδαμε ότι η απάντηση εξακολουθεί να είναι λυπή στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, τα συμμετέχοντα μέλη αποτελούν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Όμω, ε, είναι στη μειοψηφία των μελών του ΠΟΕ, έτσι Πολλέ αναπτυσσόμενε χώρε επομένω δεν συμμετέχουν. Ποιε θα είναι οι συνέπειε στι χώρε αυτέ και ποιε θα είναι οι παγκόσμιε συνέπειε αν ε, επιτευχθεί η συμφωνία. Και δεύτερη ερώτηση που αφορά επίση στην Κίνα. Οι Κινέζοι εκπρόσωποι αναφέρουν ε, ότι προσπαθούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογή των διαπραγματεύσεων ποια είναι η στάση της Κίνας σήμερα. Και βλέπετε την Κίνα ως το μεγαλύτερο κίνδυνο ότι μπορεί πιθανόν να μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χάντσεν. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για τη διαφορά μεταξύ των προσωπικών δεδομένων και των μη προσωπικών δεδομένων. Γιατί διαπιστώνουμε ότι για τα προσωπικά δεδομένα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ροών και μεγάλο πρόβλημα αποδοχής και προχωράμε πάρα πολύ αργά για να μην μπούμε καθόλου. Δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για τα μη προσωπικά δεδομένα ακριβώς να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο θέμα αυτό, γιατί λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε το μοντέλο μας και να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Ξέρω όμως ότι η Κομισιόν θα μου πει θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων. Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να ξεκινήσουμε τις εργασίες ε, από αυτές τις διαφοροποίησεις και από αυτού του ορισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you, Σόλτς. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για τη λεπτομερή παρουσίαση. Πιθανότατα κανείς δεν υποτιμά τη σημασία των διαπραγματεύσεων αυτών μια τέτοια συμφωνία σε του ΠΟΕ. Γιατί σε όλες τις χώρες θα τίθεται προκλήσεις ε, από το μέλλον του εμπορίου και συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλω καταρχήν να ρωτήσω πόσο μακριά στις διαπραγματεύσει έχετε φτάσει για να θέσετε ως προτεραιότητα ότι αυτό το δεστό εμπόριο εξυπηρετεί το συμφέρον των κοινοτήτων, των κρατών, των δήμων της τοπικής αυτοδίκησης, γιατί πρέπει να εγγυηθούμε την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα για όλους, για να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη. Να μην υπάρχει λοιπόν ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε προς τα που θα πάμε. Δεύτερον, αναφεραίνεται ότι για τον επόμενο γύρο θα υπάρχει το πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Ε, ξέρω ότι έχουμε τους ε, ραδιοτηλεοπτικές ε, εταιρείε που φύγονται από το θέμα της μεταφοράς των δεδομένων. Γιατί σήμερα αυτό θεωρείται μέρος της εμπορικής ροής, των εμπορικών ροών. Αυτό σημαίνει ότι οι διατηλεοπτικές εταιρείε τα κανάλια θα πρέπει να καλύψουν το θέμα. Και πόσο μακριά αυτό το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών ραδιοφωνικών σταθμών ε, είναι εγγυμένο, δηλαδή ότι θα εξυπηρετήσουν το συμφέρον των κοινοτήτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καλυφθεί ως ένα ειδικό θέμα των διαπραγματεύσεων. Και τέλος, Πώς ε, θέλετε να διευκολύνετε την πρόσβαση για τη δυνατότητα πρόσβαση στα ενδικά μέσα, σε περίπτωση που υπάρχουν ε, διαφωνίες. Θα έλεγα να έχουμε και μια κρόση κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ευρύ το θέμα που συζητούμε. Και ελπίζω να καλύπτεται και η ανθρώπινη νοημοσύνη, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Χαουτάλε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πραγματικά συγχυστικό. Μιλάμε για τη Συμφωνία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ στην πραγματικότητα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα ζητήματα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σχεδόν και όλους τους ψηφιακούς ε, κανόνες που απαιτούνται, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα από τις χώρες. Και κατόπιν ερχόμαστε στο σημαντικό και σχεδόν επικίνδυνο θέμα, το ownership. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες όπως η Κίνα κινούνται προς ε, ένα πλήρες ε, ownership ε, στην νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια και όταν συζητήσαμε την συμφωνία με τη Βιετνάμ είδαμε ότι το κινέζικο μοντέλο του νόμου για την κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ίσως, όχι το μόνο, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη της συμφωνίας και την ε, κύρωση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Αποτελεί μεγάλο εμποδίο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αν ε, δεν ε, μπορούν να είναι βέβαιες ότι είναι ασφαλή τα δεδομένα στη χώρα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ζητήσουμε διαφάνεια και προδραστική δέσμευση από τους νομοθέτες αλλά και τους πολίτες όλοι θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις ε, και να τους διαβουλεύονται και να μπορούν να συνεισφέρουν. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι, πιστεύουμε, ότι οι εμπορικέ συμφωνίες δεν είναι τα κατάλληλα βήματα για να αντιμετωπίσουμε κάθε πτυχή της ε, ψηφιακής πολιτικής. Υπάρχουν πτυχές ε, που, όπως το δίκτυο των πραγμάτων, τεχνητή νοημοσύνη και βρονασφάλεια που δεν αρμόζουν. Είναι σημαντικές λοιπόν, αλλά κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να αριθμιστούν στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών, ιδίω όταν ε, η εγχώρια νομοθεσία εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτήν την ε, ευρή ανασκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων Πολλοί μίλησαν για τα δεδομένα και τις ροές τους που ε, κατηγοριοποιούνται ιδιωτικά ή δημόσια. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τις τωρινές διαπραγματευτικές θέσεις των χωρών για τα, την ροή, τον εντοπισμό των δεδομένων, την Ιαπωνική πρωτοβουλία, ε, Πού βρίσκονται, τι θέσεις παίρνουν οι άλλες χώρες. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις όπως βλέπετε κύριε Κίνο. Έχετε 7 λεπτά. πολύ περισσότερα από 7 λεπτά θα χρειαζόντουσαν για να τεθεί ερώτηση, πόσο μάλλον να δοθεί απάντηση. Πάντως επαναλαμβάνω ότι από πλευράς Κομισιόν εμείς περιμένουμε να συμμετέχουμε στην ε, διαδικασία παρακολούθησης και εκεί θα θέσουμε και πολλά θέματα. Η δυνατότητα να ολοκληρώσουμε μέσα στην προθεσμία ε, μπορεί κάποια αποτελέσματα να τα έχουμε, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Πλήρη συμφωνία επί όλων των θεμάτων δεν είναι ρεαλιστική προοπτική, δεν έχουμε χρόνο και πρακτικά να συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Πολλοί συνάδελφοι ρώτησαν για τις ροές δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Θα προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, ε, τα προηγούμενα τρία χρόνια παρουσίασε ενοποιημένη ενιαία θέση για αυτό το σύνθετο θέμα αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ ροής, εντοπισμού από τη μια και ιδιωτικότητας από την άλλη. Όταν αναπτύσσαμε την προσέγγιση μας, τότε άρχισε το GDP να εφαρμόζεται πλήρως. Αυτό λοιπόν το προσέξαμε ιδιαίτερα. Και μετά διαμορφώθηκε νέα θέση η οποία παρουσιάστηκε σε κάθε διαπραγμάτευση γιατί προκειμένου περί θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορεί να έχουμε ε, με την Αυστραλία άλλη θέση όταν διαπραγματευόμαστε τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και άλλη με άλλη χώρα. Εμείς θέλουμε να επικεντρώσουμε τις ε, πειθαρχίες, τις ρυθμίσεις στα προβλήματα που έχουν σημασία για την οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα. Τα βασικά εμπόδια για το εμπόδιο είναι στον τομέα του εντοπισμού των δεδομένων. Οι προτάσεις μας λοιπόν εστιάζουν εκεί ακριβώς. Παράλληλα όμως, για να διασφαλίσουμε ότι τα, μέλη, τα μέρη ή τα μέλη ε, θα μπορέσουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητα στο επιθυμητό από εκείνους επίπεδο, γιατί η Κομισιόν συμφωνεί με όλους από εσά που μας υπενθυμίσατε ότι ο ΠΟΕ δεν είναι οργανισμός προτυποποίησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει εκεί για να αποφασίσει ποιο επίπεδο ιδιωτικότητας θα επιβάλλουν τα μέλη. Ο ΠΟΕ θέλει να διασφαλίσει ότι κάποιες βασικές αρχές ε, θα τύχουν σεβασμού, αλλά τα μη εμπορικά θέματα αυτά θα πρέπει να ε, αποφασίζονται. Αυτό αφορά και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ε, ιδιωτικότητα κλπ. Για να μπορούν τα μέλη λοιπόν να διατηρούν την δυνατότητά τους να αποφασίζουν για την ιδιωτικότητα, χρειάζονται ρυθμίσεις ή πειθαρχίες που θα ε, συνάδουν με μία ε, ε, εξαίρεση που θα είναι ευρύτερη από αυτή που υπάρχει στον, στο, στις ρυθμίσεις του ΠΟΕ. Τέθηκαν κάποιες φιλόδοξες προτάσεις όπου η ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων είναι το πρώτο θέμα, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη εξαίρεση για όλα τα άλλα, ε, εκτός από την ιδιωτικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση στην ε, εναρκτήρια φάση των διαπραγματεύσεων. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για τις ροές δεδομένων, γιατί η συζήτηση στο τέλος του Οκτωβρίου δεν θα επιτρέψει να μπούμε σε βάθος στα θέματα. Θα διευκρινίσουμε τις θέσεις μας, αλλά αν επρόκειτο να διευκρινίσω ένα θέμα το οποίο θα είναι το βασικό, μάλλον θα είναι οι ροές των δεδομένων. Οπότε θα έχουμε χρόνο για να μπούμε στις λεπτομέρειες. Τώρα, η κινέζικη πρώτα, έγγραφη πρόταση είναι πολύ προκαταρκτική έχει να κάνει με τη διευκόλυνση των ε, δασμολογικές διευκολύνσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές και τα συναφή, ε, θέματα logistics ε, και σχετικές υπηρεσίες ή μη διάκριση της υποδομής των τηλεπικοινωνιών, εταιρείε που κάνουν εμπόριο αγαθών. Αυτά είναι τα ευρύτερα θέματα πέρα από τα στενά εμπορικά. Θα χρειαστούν χρόνο όλα αυτά, αλλά είναι μια σημαντική πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις. Αρχικά υπέβαλαν τις προτάσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, στη Γενέβη δεν συζητήθηκαν καθόλου. Θα αρχίσουν να συζητιούνται τα θέματα τα δασμολογικά ε, στο τέλος Οκτωβρίου. Τώρα, για την ε, ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις ε, στην πρόταση επιτάπητος για τις μικρομήμιε, αλλά υπάρχει ένας λόγος. Ο ψηφ... ψηφιακό εμπόριο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, κάθε αυτά, είναι πύλη για καλύτερη ολοκλήρωση των ΜΜΕ στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί παρακάμπτουν έτσι όλοι οι περιορισμοί υποδομών που αντιμετωπίζουν συνήθως οι μικρές επιχειρήσεις ε, μέσα από το ψηφιακό εμπόριο μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξορισμού λοιπόν η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι το λέμε εμείς στον ΠΟΕ, η ψηφιακού εμπορίου θα ε, ωφελήσει ιδιαίτερα τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ ισχυρό αυτό εργαλείο δυνητικά για να παρακάμψουν τους περιορισμούς που έχουν συνήθως όταν θέλουν να κάνουν εξαγωγές. Αν θέλουν να εξάγουν, ας πούμε, από τη Νότια Αφρική πουλερικά, έχουν πολλούς περιορισμούς. Ενώ το ψηφιακό εμπόριο επιτρέπει σε μικρές χώρες ε, ε, και μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Η κινέζικη πολιτική για τα δεδομένα, τη ροή τους, το εντοπισμό, ε, αναγνώριση προσώπου και πράγματα που είναι ιδιωτικά. Αυτό είναι μία πρόκληση. Η Κίνα προς το παρόν δεν έχει μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις, κάθε άλλο. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, το είπαν αυτό, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις κόκκινες γραμμές της. Μίλησα για την μη διάκριση των ε, ψηφιακών προϊόντων. Επίσης συμμετέχουν πάρα πολλοί ε, ειλικρινά στις ε, συζητήσεις μέχρι τώρα. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξουν οι εντάσεις με τις ΙΠΑ. Σημείωσα τα σχόλια του κυρίου Σόλτς για το δημόσιο συμφέρον που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις όταν πρόκειται για πρόσβαση δεδομένων. Έχουμε προτάσεις, τις έχουμε κάνει. Επίσης, ε, ε, η τηλεοπτική σταθμή και κανόνες τηλεπικοινωνιών. Σήμερα το διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο μέσο τηλεπικοινωνιών. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να ξαναδούμε το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και να διευκολύνουμε τη ζωή και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτές τις online ε, υπηρεσίες για να παρέχουν τις δικές τους. Η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα δεν έχει καλυφθεί ε, ως τέτοια, αλλά σίγουρα θα προωθηθεί ε, εμέσως, αλλά δεν έχουμε θέμα που να ονομάζεται έτσι. Είναι μεγάλο μια μεγάλη πρόκληση. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο όλες τις προτάσεις της. η κοινή γνώμη έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ε, έχουμε συμμετάσχει σε διαλόγους με την κοινωνία των πολιτών για τις ροές των δεδομένων και οπωσδήποτε αυτό είναι ένα θέμα που θα συνεχίσουμε να θέτουμε με τους εμπλεκόμενους ε, πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και ο ιδιωτικό τομέα έχουν πρόσβαση και ποτέ δεν απέρριψα αιτήματα για συναντήσεις. Και βέβαια συμφωνώ με την άποψη ότι ο... μη εμπορικά θέματα δεν συζητούνται στον ΠΟΕΔΑ και δεν πρέπει. Ευχαριστώ, εισηγητή. Ευχαριστώ πραγματικά για όλες αυτές τις σκέψεις. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Είναι πολύ ε, ε, πυκνό το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα έρθουμε σε επαφή για να ξεκινήσουμε τις εργασίες στην ομάδα εργασίας για να παρακολουθήσουμε από κοντά εκ του σύνεγγυς αυτές τις διαπραγματεύσεις. Sure Βεβαίω. Και είμαι σίγουρο ότι θα παρακολουθούμε πραγματικά από κοντά αυτέ τι διαπραγματεύσει γιατί είναι κοινού μα ενδιαφέροντο. Αυτό κλείνει αυτή τη συζήτηση. Έχουμε τώρα το σημείο 10 για την ε, αλλά τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για τα πουλερικά. Υπήρξε μια αύξηση κρέατος πουλερικών ξαφνικά και άρα το ερώτημα είναι πού βασίζεται αυτή η αύξηση και ποια είναι η ε, δασμολογική κατάταξη. Έκανε μία πρόταση τώρα η Κομισιόν. Ε, η κυρία Κλάρκ, πολύ γνωστή από την αρμόδια ο κύριο Κλάρκ, συγγνώμη, τη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν, θα μας κάνει μια παρουσίαση για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω πολύ λιγότερο από πέντε λεπτά. Ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας υπάρχει μια ε, ευρύτερη του περιεχομένου εμπορική συμφωνία, ε, από την οποία αποφελούνται και οι δύο πλευρές. Υπήρχε όμως μια εξαίρεση ε, ο τομέας των πουλερικών δεν απελευθερώθηκε, είναι ευαίσθητος τομέας. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί για την απελευθέρωση, προσφέρουμε στην Ουκρανία ε, μια ποσόστοση 20.000 τόνου πουλερικών και δύο στήθου πουλερικών. Από το 2016 παρατηρήσαμε μια αύξηση στι εξαγωγέ από την Ουκρανία στήθου πουλερικών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4.000 τόνους το 2016, 27.000 τόνοι το 2017 και 55.000 τόνοι περίπου το 2018 φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμία ή μια, ένα παραθυράκι στην ε, ε, συμφωνία. Υπήρχαν άλλες απελευθερωμένες δασμολογικές κλάσεις ε, μέσω των οποίων μπορούσαν να εξάγουν υψηλής ποιότητας κρέας στήθους πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να παρακάμπτουν συμφωνία. Είναι κάτι το απόλυτα νόμιμο. Το στήθος των πουλερικών όμως, τα προϊόντα αυτά και τα πουλερικά γενικά είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία για, την, για τα, Ευρω... για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπραγματευτήκαμε λοιπόν με την Ουκρανία για να μπει ένα τέλος σε αυτή την διαφορετικά ε, ατέλειωτη αύξηση ε, των εισαγωγών αυτών Πρόσφατα συμφωνήσαμε με την Ουκρανία ότι θα υπάρξει ένα όριο ε, στις 50.000 τόνους για τις εξαγωγές αυτές ε, στήθους πουλερικών και ταυτόχρονα θα κλείσουμε και το παραθυράκι που υπήρχε στη συμφωνία. Αυτή, αυτό λέει το σχέδιο συμφωνίας που έχετε ενώπιόν σας. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σας ε, ειδοποίησαμε, Πρόεδρε, ότι επιθυμούμε να ε, εφαρμόσουμε τη συμφωνία αυτή σε προσωρινή βάση, αναμένοντας την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λόγω του πόσο επίγονη ήταν να αναχαιριστούν αυτές οι εισαγωγές από την Ουκρανία. Κατά τη γνώμη μας η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη. Η Ουκρανία δέχεται το όριο αυτό στις εξαγωγές της πουλερικών προς την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύοντα και τους ε, παραγωγούς της. Ε, διαφορετικά, χωρί αυτή τη συμφωνία, η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να εξαγάγει απεριόριστες ποσότητες αυτού του προϊόντος. Έχετε, έχει, όπως ξέρετε, η Ουκρανία μεγάλη δυναμικότητα παραγωγής στον τομέα αυτό. Αυτό το όριο λοιπόν των 50.000 τόνων θα προστατεύσει ε, τον εγχώριο τομέα πουλερικών. Αναμένουμε η Ουκρανία να ε, επικυρώσει τη συμφωνία αυτή τον Νοέμβριο και γι' αυτό θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή Ίντα να κινηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα από την πλευρά της για να ε, τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Η μόνιμη εισηγήτρια έχει το λόγο. Κύριε Γκιώρη. ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενημέρωση και που μας παρουσίασε και το πλαίσιο του ζητήματος. Αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, για να σας διασκεδάσω θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου για να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Όταν ε, πρώτο άκουσα ε, την υπόθεση αυτή, τότε σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή στο να το κάνω αυτό. Δηλαδή να αφήσουμε ένα παραθυράκι, τότε αυτοί το χρησιμοποιούν. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και αναμφισβήτητα είναι πολύ σημαντικό εταίρο η Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατηγικά, αλλά προφανώς είναι προς το συμφέρον μας. να έχουμε ως δυνατόν περισσότερες εμπορικές συμφωνίες μαζί τους. Αλλά είπα, αν υπάρχει κάποιο παραθυράκι, τότε ο άλλος εταίρος θα χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θέλω να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να προσπαθήσει να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια. Γιατί ας μην είμαστε ανόητοι, γιατί αν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες κάποιος πάντοτε τις εκμεταλλεύεται. Ιδίως δεν μπορούμε να αφήνουμε τρίτες χώρες να μπαίνουν ε, με αυτόν τον τρόπο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε μπορούμε να θέτουμε σε δυσκολία τους αγρότες μας για τέτοιους λόγους. Αν έχουμε μια συμφωνία μάλιστα πρέπει να την εφαρμόσουμε. Προφανώς ε, η ερώτηση είναι πώς χρησιμοποιούμε τις συμφωνίες αυτές και πώς παρατηρούμε Πώ ελέγχουμε την εφαρμογή των συμφωνιών. Θέλω λοιπόν να ζητήσω την Κομισιόν να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Και όταν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την εφαρμογή της. Νομίζω ότι είναι καλή η λύση αυτή, την υποστηρίζω. Φαίνεται ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να τη δεκτεί γιατί είναι πολύ σημαντική και για τα δύο μέρη. Αλλά έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, θα μπορούσε ε, η Κομισιόν να βρει αν υπάρχουν και άλλα παραθυράκια σε άλλες συμφωνίες, παραδείγματο χάρη. Και δεύτερη ερώτηση. Η Κομισιόν δεν είχε σκεφτεί να παρακολουθήσει έχει σκεφτεί να παρακολουθήσει τη συμφωνία αυτή, να υπάρχει μια συνέχεια δηλαδή. Ο κύριος Μπέλκα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η Κομισιόν επαναδιαπραγματεύτηκε μια δεσμολογική συμφωνία με την Ουκρανία. Κλείνει έτσι το παραθυράκι, στο οποίο μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι παραγωγή στήθους πουλερικών της Ουκρανίας. Θεωρήθηκε ευαίσθητο το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών. Όμως λυπούμαστε που ως μέρος της ε, τροποποίησης των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πληρικών ο όγκος της ποσόστοσης ε, θα αυξηθεί σημαντικά. Δηλαδή από τις 20.000 ε, θα πάμε στις 70, πάνω από τρεις φορές. Φυσικά αυτό ανησυχεί τους Ευρωπαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Επίσης θέλω να επαναλάβω την ερώτηση που έθεσε η προλαλήσασα. Πώς αξιολογούμε αυτή την κακή εμπειρία αυτού του μέρους της συμφωνίας. Πώς θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Πώς θα το παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ID δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σολτζή Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους του σκιώδου συζητητού μας που δεν είναι εδώ σήμερα. Θέλω να τονίσω ότι προφανώς είναι πολύ ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα. Και παρά το μέγεθος των εισαγωγών και των εξαγωγών, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο θέμα της ευμερίας των ζώων και αν υπάρχει σχετική εγγύηση στην Ουκρανία και κατά την παραγωγή του κρέατος αλλά και κατά τη μεταφορά αν έχουμε ζωντανά κοτόπουλα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνδέεται επίσης με το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Περιλαμβάνονται τώρα αρκετά στο κείμενο της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σροϊερ Πιέρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από το Βέλγιο και τις κάτω χώρες για το θέμα αυτό από πέρσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση αυτή. Και από το 2018 πολλοί ένωσαν τη δυνάμει του. Υπάρχει εδώ ένα νομικό κενό στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, αναφεσβήτητα, αλλά δεν αρκούν οι τροποποιήσεις, γιατί τελικά ε, επικροτείται και ανταμείβεται η κακή συμπεριφορά. Δεν είναι ίσονο σημασία στο ζήτημα αυτό. Επίσης, ταυτόχρονα είναι σημαντικό να σταματήσουμε αυτή την ε, εισρωή φτηνού ε, στήθος κοτόπουλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ουκρανία. Αυτό είναι εις βάρος των γεωργών γιατί ε, αναγκάζονται να παράγουν με πολύ ψηλότερο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, ναι, είμαστε υπέρ των αλλαγών, αλλά δεν είναι ιδανική η λύση και η Ουκρανία ε, δεν της αξίζει να σωθεί η υπόλοιψή τη. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τι συμβαίνει και ο Ολλανδικός τομέας των πουλερικών λέει ότι τουλάχιστον είναι καλύτερο από το τίποτα. Επόμενη μιλήτρια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και από τη σκοπιά της ε, ευημερία των ζώων θέλουμε να τονίσουμε εμείς. Υπάρχουν βέβαια και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά. Το κόστος ε, παραγωγής των πουλερικών στην Ουκρανία είναι 22 φορές χαμηλότερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Ουκρανία δεν φαίνεται, πάντοτε δεν φαίνεται να σέβεται απαραίτητα τις δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά την ε, κτηνοτροφία πουλερικών σε βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις και ε, έχω και κάτι άλλο. Ε, τη στιγμή που έχουμε ε, κλιματικές φιλοδοξίες και στόχους που πρέπει να πετύχουμε, θα έπρεπε επίσης να σκεφτούμε από κοινού να διαδώσουμε το δικό μας μοντέλο και να θέσουμε το ερώτημα αν είναι σκόπιμο να αυξάνουμε τις εισαγωγές πουλερικών όταν ε, μιλάμε ε, για κτηνοτροφία που ε, μπορεί να λάβει χώρα και αλλού. Και τα ίδια φυσικά αφορούν και τις συμφωνίες με τη Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ από την Επιτροπή Γεωργίας. Έχουμε τον κύριο Κουτσμίκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή Γεωργίας υποστηρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής και είναι υπέρ της ε, ταχύτερης εφαρμογής της μέσω της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας ε, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναγωγών για τα προϊόντα πουλερικών. Πρέπει να ε, σταματήσουμε τη δυνατότητα να εισαγάγουμε περισσότερα τέτοια ε, τεμάχια ε, που δεν σέβονται τα πρότυμα. Έχουμε φτάσει στους 55.000 τόνους το 2018, δηλαδή είχαμε 15 φορές αύξηση από το 2016. Η εισαγωγή αυτών των στήθων με τα βραχίωνα από έχει δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα στην αγορά πουλερικών προκαλεί ανισορροπίες ε, στην αγορά. Η Επιτροπή Γεωργίας ε, θα ήθελε να τονίσει τρεις σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και ελπίζουμε να τις σημειώσει η Κομισιόν. Καταρχήν, αν συμφωνία τεθεί σε εφαρμογή, θα θέλαμε να αλλάξουμε τη δεσμολογική ποσόσταση και να έχουμε μονομένε δεσμολογικέ γραμμέ και να τι παρακολουθούμε ένα μήνα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αλλάξει αμέσω τα πράγματα για να αποσταθεροποιήσει την ευρωπαϊκή αγορά πουλερικών και ιδίως την πολωνική αγορά. Γιατί ε, μέσω της Πολωνίας περνάνε αυτές οι εισαγωγές κυρίως. Δεύτερον, προτείνουμε να προτείνει η Κομισιόν στην Ουκρανία να τροποποιηθεί η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, θα πρέπει να ε, εισαχθούν διμερείς, ε, μάλλον προστασία, διμερείς για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να αλλάξουν τις ασμολογικές ποσοστώσεις αν υπάρχουν διαταραχές σε ευαίσθητους τομείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχετε μια εισαγωγή από την Ουκρανία που αποσταθροποιεί τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών θα πρέπει να ε, περιλαμβάνει ένα μηχανισμό που να επιτρέπει την ε, αυτόματη εμπλοκή. Και τρίτον, θα πρέπει να δεσμεύσουμε τους Ουκρανούς εταίρους μας, να διασφαλίσουμε ότι θα σέβονται τους υγειονομικούς και φυτογειονομικούς κανόνες, καθώς και τις διατάξεις για την ευημερία των ζώων. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστά τα πρότυπα. Επομένως, η Επιτροπή Γεωργίας είναι υπέρ της συμφωνίας αυτής, αλλά θέλουμε αυτές οι τρεις προϋποθέσεις που σας ανέφερα να είναι μέρος της συμφωνίας. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, βουλευτές που σχολίασαν με ερωτήσεις. Να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε θέμα. Καταρχήν ρωτήσατε αν το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει και σε άλλες ε, συμφωνίες ΣΕΣ. Όχι εξετάσαμε προσεκτικά κάθε υπάρχουσα και μελλοντική Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών και αυτό το κενό δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί να υπάρχει, οπότε να είστε βέβαιοι πάνω σε αυτό. Δεύτερον, η παρακολούθηση και η εφαρμογή από την Ουκρανία της ρύθμισης αυτής. Χάρη στην πολύ στενή παρακολούθηση εντοπίσαμε καταρχήν το θέμα νωρίς και η Ουκρανία πρέπει να παρουσιάσει στα τελωνία στην Ευρώπη μια δήλωση καταγωγής, πιστοποιητικό που θα δείχνει ότι μπορεί να ε, ευνοηθεί από την προτιμησιακή δασμολογική ε, κλάση και δεν ανησυχώ. Προφανώς και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πιστή εφαρμογή αυτού της νέας ρύθμισης ε, ποσόστοσης από την Ουκρανία. Ο όγκος είναι σημαντικός, περίπου 50.000 τόνοι, αλλά, όπως είπε ένας συνάδελφος, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δίνουμε πρόσθετο όγκο στην Ουκρανία, λιγότερο όμως από ό,τι εξήγαγε πέρσι. Οπότε νομίζω ότι ε, βάλαμε ένα αποτελεσματικό ανώτατο όριο στον όγκο και δεν θα αποσταθοεροποιηθεί ούτε θα διαταραχθεί η ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι η τάξη μεγέθους ανά, τέτοια. Τώρα, για την καλή κατάσταση των ζώων, με ή χωρίς συμφωνία ΣΕΣ, η Ουκρανία, ως οποιαδήποτε εξαγωγός χώρα, θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι διαπραγματεύσιμοι μέσα από ΣΕΣ. Τώρα για την καλή υγεία των ζώων και την καλή τους κατάσταση, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερικές μέρες θα εγκρίνει ένα παράρτημα για την ε, καλή κατάσταση των ζώων που θα ενταχθεί στη Συμφωνία Ένωσης Ουκρανίας και αυτό θα εγκριθεί από την Ουκρανική πλευρά. Αυτό δεν συνιστά έναν οδικό χάρτη με πρακτές προθεσμίες καταληκτικές, ώστε να προσαρμοστεί ε, στο ενωσιακό εκτιμένο η Ουκρανία όταν πρόκειται για νομοθεσία ασφάλεια, υγεία κλπ. Η Ουκρανία θα είναι η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα, εκτός από την Ελβετία αν θέλετε, σε έναν βαθμό που προσαρμόζεται προς τους κανόνες ε, της Ένωσης για την καλή κατάσταση υγεία και ασφάλεια. Αυτό το χαιρετίζουμε. Ε, βοηθεί να υπάρχουν ίσοι κανόνες του παιχνιδιού και να εφαρμόζονται πιστά οι κανόνες μας και τα επόμενα χρόνια. Θαυμάσια. Πολύ ωραία. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ε, τις δέχομαι. Ε, το ε, άκουσα και το αίτημα της Επιτροπής Γεωργίας. Η Κομισιόν θα επανέλθει όμως οπωσδήποτε με τα, στα θέματα αυτά. Από ό,τι γνωρίζω, οι υγειονομικοί, φυτογειονομικοί κανόνες συμπεριλαμβάνονται και στην Αρχική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, οπότε οι προϋποθέσεις υπάρχουν και τονίζω πάλι τη σημασία της παρακολούθησης και επαγρύπνησης για τα θέματα της εφαρμογής της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Οπότε γρήγορα καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα και η συγγήτρια και οι Σκιώδης θα προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν αφού δεν υπάρχει άλλωστε και καμία αντίρρηση στη συμφωνία αυτή. με τις προϋποθέσεις βέβαια που έθεσε και η Επιτροπή Γεωργίας. Εντάξει, οπότε τελειώσαμε το σημείο 10 και προχωρούμε στο σημείο 11. Και τώρα αλλάζω καπέλο και γίνομαι μόνιμος εισηγητής για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πριν από 10 χρόνια ε, συνήψαμε μία συμφωνία μια συνεννόηση ε, με βάση τη συνεχιζόμενη συζήτηση για την εισαγωγή βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σαφή δέσμευση προς τους καταναλωτές να μην επιτρέψουμε εισαγωγές βοήου κρέατος που θα αντιμετωπίζεται με ορμόνες. Έχουμε απαγορεύσει βόηο κρέας με ορμόνες όπου ε, και ο Κόντεξ Αλιμεντάριους έχουν άλλη γνώμη. Γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν πορίσματα επαρκώς επιστημονικά ότι το ε, βόλιο κρέας με ορμόνες ε, θα υποσκάψει την ανθρώπινη υγεία. Εμείς όμως τις αρχές μας τις στηρούμε. Και Κάποιες χώρες που ε, παράγουν βόλιο κρέας ε, έθεσαν ζήτημα. Βρέθηκε μια συμφωνία. επιτρέπομε 45.000 ε, τόνους υψηλής ποιότητας βοήου κρέατος, αυτή την η να εισάγεται αλλά χωρίς ορμόνες. μετά τις συζητήσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε και συγκεκριμένα μετά τη συνάντηση Juncker-Trump έγινε μια συζήτηση για την ποσόστοση αυτή που βέβαια ήταν ως προς το μεγαλύτερό της μέρος προς τις ΗΠΑ. 45.000 αυτό χωρίστηκε μεταξύ ΗΠΑ, Αυστραλία, Ουρουγουάι και Αργεντινή. Και ε, δόθηκε υπόσχεση να δοθεί μεγάλο κομμάτι στη ΣΥΠΑ. Η πρόταση είναι να δώσουμε 35.000 τόνους από τις 45.000 συνολική ποσόστοση. 35.000 να δοθούν στη ΣΥΠΑ. Ευτυχώς η Αυστραλία, η Ουρουάη και η Αργεντινή συμφωνούν με την πρόταση αυτή παρόλο που αυτό σημαίνει ότι μειώνουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες στα πλαίσια αυτής της ποσόστοσης, δηλαδή χωρίς δασμούς. Δεν είμαι βέβαιος τι έδωσε η ή κάποιος άλλος στις χώρες αυτές για να συμφωνήσουν. Εν πάση περιπτώσει συμφώνησαν με την ποσόστοση αυτή. Εμένα είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Είναι ένα άλλο βήμα προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ μετά τη συναντηση Γιούγκερ Τραμπ. Εισαγάγαμε περισσότερους ε, σπόρους σόγιας μετά από τη συνάντηση, περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Προχωρούμε με προτάσεις αλλά και κάνουμε βήματα υπέρ των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού βλέπουμε ότι δασμοί στο χάλιβα υπάρχουν για τον αλουμίνιο επίσης. Για τα καρτέλ επίσης υπάρχει η απειλή για, τα, για άλλα προϊόντα υφίσταται. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Έχουμε ένα θέμα με τα, τις ελιές τις ε, ισπανικές και τώρα θα μάθουμε και νεότερα για το Airbus και τους έξτρα δασμούς από τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι έχει εκδοθεί η απόφαση και σύντομα θα ακούσουμε και για τα μέτρα. Και αυτά είναι μόνο η αρχή του καταλόγου σε σχέση με τις ενέργειες των ΙΠΑ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το μικρό ζήτημα του βοήου κρέατος έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη στάση απέναντι στη ΣΥΠΑ, ότι ναι, να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις, ε, αφού από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν έχουμε δει ούτε μία κίνηση προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης. Οπότε υπάρχει πλήρης απουσία ανάληψης δράσης από αμερικανικής πλευράς. Παρ' όλα αυτά είμαι ανοιχτός στη συζήτηση που θα ακολουθήσει για την πρόταση αυτή δεν θα βλάψει τους παραγωγούς γιατί η ποσόστοση δεν αλλάζει απλώς δίνουμε ένα μήνυμα προς τις ΙΠΑ λέμε ότι ε, ε, θέλουμε να τηρήσουμε τους κανόνες θέλουμε όμως και να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση και τώρα δίνω το λόγο στον Σκιώδη και ξαναγίνομαι πρόεδρος Ποιος θα μιλήσει? Ο κύριος Χάνζεν. Ευχαριστώ πολύ, Μπέρντ. Ακόμα δεν είμαι επίσημα σκιώδης, ως, δεν είμαι σκιώδης, ως συντονιστής αναλαμβάνω σήμερα, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε πρώτα τους συναδέλφους και να γίνει ε, η ανάληψη ας πούμε, των καθηκόντων. Μου φαίνεται ότι Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοιτάω και την ώρα. Περιμένουμε το, την απόφαση από τον ΠΟΕ για την υπόθεση Airbus. Τα επόμενα λεπτά πρόκειται να ληφθεί η απόφαση. Δεν την έχω λάβει ακόμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι να δούμε τι θα γίνει, ε, τι θα προσφέρουν και εκείνοι Επίσης σήμερα το πρωί είχαμε εδώ Αυστραλιανή αντιπροσωπεία από μια χώρα η οποία θέλει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Η Αυστραλία θα ε, παίξει ρόλο. Γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Χρόνος υπάρχει και δεν χρειάζεται να ε, παραδώσουμε όλα μας ε, τα όπλα από τώρα. Ε, ας αφήσουμε και ένα διαπραγματευτικό ατού για, ε, για την Επιτροπή, για να διαπραγματευτεί υπέρ των θέσεών μας. Από το Ρινιού... Ευχαριστώ. Στείλαμε μια επιστολή στο Κογκρέσο αυτή τη βδομάδα εξ ονόματος αρκετών συναδέλφων εδώ και με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω που προσυπογράψατε. Πολλοί ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες και κράτη-μέλη ε, ε, πολλοί υπέγραψαν. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία για τα διατλαντικά θέματα. Καλούμε το Κογκρέσο σε αυτή την επιστολή να εργαστεί μαζί μας ε, ώστε να ε, μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ιδιαίτερα και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ σε σχέση με τη συμφωνία του 2018 που θα αναφέρουμε αργότερα ακολουθήσαμε πολύ επικοδομητική στάση, ελπίζουμε ότι οι θα κάνουν το ίδιο. Τώρα, αυτό για το βόλιο κρέας χωρίς ορμόνες, ακούσαμε ότι η Αυστραλία απογοητεύτηκε γιατί μειώθηκε το δικό της το μερίδιο, αλλά αναρωτιέμαι, οι άλλοι εταίροι τι είπαν, πώς αντέδρασαν, δηλαδή μειώνουν τις ποσοστώσεις, αλλά δεν θα κάνουν εξαγωγές τόσο πολλές όσο έκαναν μέχρι τώρα. Και επίσης οι σχέσεις μας, οι εμπορικές μαζί με τις χώρες αυτές, ε, πώς θα επηρεαστούν από όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόφερ δεν είναι εδώ. Ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για την, το, προβληματική, τη γενικότερη. Τώρα πώς η κοινή δήλωση αυτή πώς θα εφαρμοστεί. Ε, θα περιοριστώ σε δύο παρατηρήσεις. Τι συνέχεια θα δοθεί στην κοινή γεωργική πολιτική. Η Ιρλανδία θα πρέπει να, ε, πάρει, ε, να έχει υποστήριξη, ούτως ώστε να ε, αναδιοργανωθεί και πρέπει να δούμε και τις αγωγές. Επίσης, η ουδετερότητα του κλίματος, η δικαιοσύνη σε θέματα αλλαγής κλίματος, όλα αυτά που επηρεάζουν σήμερα θα πρέπει να συζητηθούν και η το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα που αφορά μια συμφωνία θα πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό έχει νόημα να κάνουμε αυτές τις εισαγωγές και ρωτώ εδώ την Κομισιόν αν παράλληλα ε, θα πρέπει ενδεχομένως να κλείσουμε μια, ε, κάποιες μονάδες παραγωγής. Ο κύριος Μπουζά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζουμε το σημείο 11. Είναι μια ε, θετική πρωτοβουλία για ε, να διευρυνθούν οι διατλαντικές συνομιλίες. Νομίζω ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας τα προβλήματα που προέκυψαν με τους δασμούς ε, για το χάλιβα και το αλουμίνιο, που επηρεάζουν ε, μια σειρά από βιομηχανικά προϊόντα. Ε, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας ενώ ε, παράλληλα θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Και μάλιστα θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να έρθει και να κάνει μια επεξηγηματική δήλωση στην ε, ε, Επιτροπή Παρακολούθησης, γιατί εμπλέκονται τόσο πολλά συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις αυτές με τις ΗΠΑ. Και ένα βασικό παράδειγμα είναι η υπόθεση του Airbus, που σημαίνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα υιοθετήσουν κάποια μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε με τη σειρά να πάρει μέτρα ε, λόγω των, ε, του Boeing, πράγμα το οποίο δεν θα βοηθήσει καθόλου τον διατλαντικό διάλογο αν υπάρχουν ενδείξει αύξηση των εισαγωγικών δασμών εκ μέρου των ΗΠΑ, η μόνη λύση είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε και να σταματήσουμε αυτή την καθοδική πορεία ε, προστατευτισμού μέτρων και αντιμέτρων και αντιπίνων που ε, μας οδηγεί πολύ γρήγορα στον κατήφορο. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι η Κομισιόν θα βρει έναν τρόπο να βγούμε από τον κίνδυνο αυτό και ταυτόχρονα, όπως είπα, θα πρότεινα η Κομισιόν να έρθει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τη νέο συσταθήσα όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση. Υπέγραψα μια ε, επιστολή μαζί με τον συναδελφό μου και λέμε ότι το κάθε τι θα ήταν καλύτερο από το να κολλήσουμε σε μια τέτοια διαμάχη. Ευχαριστώ. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή παρακολούθηση όταν όλες οι πολιτικές ομάδες θα έχουν ορίσει τους εκπροσώπους τους. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε τη συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ στην ε, Επιτροπή αυτή. Μόλις ε, βγει η απόφαση για το Airbus, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έχουν δικαίωμα σε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και έχουν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν και ότι δεν θα διαπραγματευτούν μαζί μας. Και είναι κάπως αντιφατικό. Είναι μια αντιφατική αυτή η προσέγγιση του ΠΟΕ. Αυτή είναι η απόφαση βέβαια ε, στο τελευταίο επίπεδο του ΠΟΕ. Και την απόφαση αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την παίρνουν επιλέξει, ενώ από την άλλη πλευρά του νομίσματος υπονομεύουν την πιθανότητα το σώμα αυτό προσφυγών να απορρίψει τον ορισμό, διορισμό νέων δικαστών για το σώμα αυτό. Ήταν μια σύντομη παρέμβαση αυτή, αλλά νομίζω απαραίτητη. Λοιπόν, ο κύριο Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε δεν είναι πολύ ρόδινη η εικόνα. Δυστυχώς οι σχέσεις μας δεν είναι όσο καλές θα έπρεπε να είναι. Είχαμε το σχέδιο Marshall μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια ε, ε επιδεινώνονται οι σχέσεις, δεν είναι καλή κατάσταση όπως είπαν οι συνάδελφοι. Η υπόθεση Airbus μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή σημαντικών δασμών σε προϊόντα όπως είναι τα γαλακτοκομικά, οι τσάντες, τα ενοπνευματότυποτά, το Ιρλανδικό ουίσκι παραδείγματος που εξάγεται στις ΗΠΑ και πολλά ακόμα. Και φυσικά ε, την ερχόμενη άνοιξη θα έχουμε και την απόφαση για την Boeing. Ε, όπως έκανε ο κύριος Γιούγκερ, ε, το ίδιο ελπίζουμε να κάνει και η πρόεδρος Βαντερ Λάιεν και ο Επίτροπος για το Εμπόριο, να ε, συνεχίζουν τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ, προσπαθώντας να αποκλιμακώσουν την κατάσταση και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Επίσης, για το βόλιο κρέας, δεν φαίνεται να υπάρχει μια αντίφαση από τη μια μεριά να έχουμε ένα πρόγραμμα επίγουσας ανάγκης, ένα κατεπήγον πρόγραμμα για τους παραγωγούς βοήου κρέατος λόγω των μεγάλων απολειών που έχουν υποστεί και μέρος του προγράμματος να είναι η μείωση της παραγωγής τους. Ενώ παράλληλα παίρνουμε μέτρα που αυξάνουν την παραγωγή σε άλλα μέρη. Πώς λογικά το εξηγείτε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι χρειάζεται πολλή συζήτηση και πολλά μαθηματικά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κύριε Κλάρκ, ακούσατε τη συζήτηση. Στην Επιτροπή είχατε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μία πρόσθετη παρέμβαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριο Σλάναγκαν, να αναφερθώ στο τελευταίο σχολείο του κυρίου Κέλλη για τα 15 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση στην παραγωγή και το έθεσε ο κύριος Σόλτς. Υπήρχε η επιλογή να μειωθεί η παραγωγή. Υπήρχε όμως και άλλη δυνατότητα. Και λυπάμαι που το λέω και το είπαμε και στη συνεδρίαση όταν εγώ και ένας συνάδελφος συναντήσαμε την Κομισιόν. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η Ιρλανδία θα επιλέξει την ε, μείωση και τελικά βγήκαμε αληθινοί. Είναι λυπηρό λοιπόν που κάναμε αυτή την επιλογή και λένε τώρα στους κτηνοτρόφους να καλλιεργήσουν δέντρα και ε, τελικά ε, να βοηθήσουν στην αύξηση του ε, δάσους. Όμως δυστυχώς η κυβέρνηση του κυρίου Κέιλι επέλεξε να μειώσει την παραγωγή του πιο φιλικού προς το περιβάλλον βόλιο κράτος που θα μπορούσατε να έχετε στο πιάτο σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, και εγώ είμαι από την κάτω και έχουμε και εμείς πολύ ωραίο βόλιο κρέα. Ο εκπρόσωπο Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς ε, στα εισαγωγικά σας σχόλια, είναι πάρα πολύ παλιά διένεξη αυτή στον ΠΟΕ από την εποχή του Μπιλ Κλίντον. Δεν έχει καμία σχέση με την ε, συμφωνία Τραμπ-Γιούνκερ πέρσι. Εμείς ε, είχαμε πει λοιπόν ε, με την ε, απαγόρευσή μας το κρέας ότι δεν θα αλλάξουμε ποτέ την απαγόρευσή μας για τις ορμόνες στο βοηοκρέας. Τι κάνουμε λοιπόν, αποζημιώνουμε τους Αμερικανούς με μία ποσόστοση 45.000 ε, τόνων ε, για βόλιο κρέας χωρίς ορμόνες. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τώρα, για να συνάδουμε με τους κανόνες του ΠΟΕ, αυτή η ποσοστοσία έπρεπε να ανοιχτεί και σε άλλες ε, χώρες προμηθευτές και σύν το χρόνο οι ΗΠΑ που στις αρχές έχεραν μονοπόλιο αυτών των 45.000 τόνων, Τελικά το μεριδιό τους μειώθηκε ε, λόγω συμμετοχής Αργεντινής, Ουρουγουάης, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας. Και φυσικά ήταν δυσαρεστημένοι οι Αμερικανοί με την κατάσταση αυτή είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν 120 εκατομμύρια ευρώ σε κυρώσεις ε, και αποφάσισαν να το κάνουν αλλά να πραγματευτούν την ποσόστοση μαζί μας ε, για να τους δώσουμε ένα εγγυημένο μερίδιο της συνολικής ποσόστοσης. Η συμφωνία λοιπόν την οποία πετύχαμε ε, δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 35.000 τόνους από την ναι, υφιστάμενη ποσόστοση των 45.000 τόνων και αυτή η αύξηση στις ΙΠΑ ε, ουσιαστικά μέσα σε 7 χρόνια μειώνεται σταδιακά. Τώρα είχαμε ερωτήσεις για τη στάση και των άλλων προμηθευτών. Δεν θα σας αποκρύψω ότι η Αυστραλία, η Ουρουάη και η Αργεντινή ήταν δυσαρεστημένες γιατί το μερίδιό τους για την ποσόστοση μειώνεται προ όφελο των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, συνειδητοποίησαν όμω ότι αν δεν φτάσουμε συμφωνία με τι ΗΠΑ, τότε οι ΗΠΑ ε, θα ε, επαναθέσουν τι εμπορικέ κυρώσει που του επιτρέπει ο ΠΟΕ και η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα θα υφίστατο και δεν θα είχαμε καμία ποσόστηση. Θα εξαφανιζόταν εντελώ η ποσόστοση. Αυτή την ε, επιλογή αντιμετώπιζαν. Έτσι λοιπόν ε, διστακτικά δέχτηκαν. Είπαν ότι αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα. Θέλω να τονίσω κυρίως τον κύριο Σόλτς ότι δεν υπάρχει αύξηση στις εξαγωγές του βιοκρατού στην Ευρώπη ως συνέπεια αυτής της συμφωνίας. Ήδη από το 2009 εισάγουμε 45.000 τόνους ε, βόλιου κρέατος υψηλής ποιότητας χωρίς ορμόνες, δυνάμει αυτής της ποσότητας. Ο όγκος παραμένει ο ίδιος, απλώς μάλλον πάντα καλυπτόταν ο όγκο αυτός, απλώ αυτό που αλλάζει είναι ότι θα έρχεται περισσότερο κρέα από τη ΣΥΠΑ και λιγότερο από τι άλλε τρει χώρε, αλλά δεν έχουμε διαφοροποίηση του όγκου, δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο αυτό ε, στο βόλιο κρέα ε, στην κάτω Σαξονία ή στην Ιρλανδία. Στο κρέα που παράγεται εκεί δηλαδή. Επίσης δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα πρότυπα που θα πρέπει να πληρούνται από τους εξαγωγείς που χρησιμοποιούν την ποσόστοση. Αυτό παραμένει άθικτο. Τα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια, αυτά μένουν ίδια και παράλλακτα. Και τρίτον, δεν αλλάζουμε καθόλου την απαγόρευσή μας ε, για το βόλιο κρέας ε, με ορμόνες. Όλο το κρέας που εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μην περιλαμβάνει ορμόνες και αυτή η ποσόστοση δεν αποτελεί εξαίρεση. Κατόπιν. Όπως είπα, αυτή η διένεξη είναι 20 ετής. και θα κλείσει ε, θα κλείσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους ε, τη διένεξη αυτή στον ΠΟΕ. Αν δείτε, υπάρχει στο άρθρο 4 ή 5 ότι μετά από 10 έτη, αν λειτουργεί η συμφωνία ομαλά που θα λειτουργήσει, τότε τα μέρη Τη Συμφωνίας Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοινοποιήσουν στον ΠΟΕ ότι έχει οριστικά κλείσει η διένεξη αυτή. Είναι νομίζω πολύ καλή αυτή η δέσμευση της Ηνωμένε Πολιτείε, ότι οριστικά θα ε, κλείσει αυτή η πληγή στις σχέσεις μας για πολλά χρόνια. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό το θέμα το είχαμε κρατήσει ξεχωριστό από τις διάφορες διακυμάνσεις των εμπορικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπόριο στα γεωργικά προϊόντα μπορεί μερικές φορές να είναι το θύμα των εμπορικών διαφωνιών σε άλλους τομείς. Θα μπορούσε να είναι και εδώ θύμα, όμως θέλαμε να το διατηρήσουμε εκτός της του ευρύτερου διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το εμπόριο. Είναι θετικό βήμα για τις ε, σχέσεις μας που αυτή τη στιγμή είναι κάπως ταραχώδης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και να πω ότι παρά το σκεπτικισμό σας, Πρόεδρε, μπορεί η Επιτροπή σας να προχωρήσει το συντομότερο προκειμένου να εγκριθεί αυτή η συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε οι νέες διευθετήσεις και το νέο μερίδιο της ποσόστοσης να μπορεί να ισχύσει από 1η Πρώτου 2020. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα θέσουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα το συζητήσουμε πολύ προσεκτικά. Και βέβαια μέρος του παιχνιδιού είναι και το πολιτικό σκέλος ε, στο όλο πλαίσιο των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί έχει έρθει εκπρόσωπος Κομισιόν για το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12, το οποίο είναι μια ευρύτερη οπτική των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μετά της κατόπιν της κοινή δήλωσης της 25ης Ιουλίου 2018. Πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου και περισσότερο. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε τέσσερα κύρια αποτελέσματα αυτής της ε, δυσέλιδης ε, συνεννόησης, αν θέλετε, μεταξύ Γιούγκερ και Τραμπ, απελευθέρωση των δεσμών για τα βιομηχανικά αγαθά. Θα πρέπει να προωθηθεί λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε ρυθμιστικά ζητήματα. Επίσης, συνεργασία για ενεργειακά ζητήματα και συγκεκριμένα επί του υγροποιημένου φυσικού αερίου και θα πρέπει να υπάρξει αύξηση σε ό,τι αφορά τους σπορσόγιας και η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος. και να προθεθεί μια κοινή συνεννόηση. αναμέναμε ότι αυτή η συμφωνία αφαιρεί 25% των δασμών που αφορά το 25% των δασμών ε, στη Χαλβουργία θα εξαφανιζόταν. Όμως, έχουμε κάποιες στοιχές από τον ψυχρό πόλεμο. Ο πρόεδρος μπορεί να θέσει δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και μα είπε, το σχάρι ότι ο Χαλίβα και το Λουμίνο που από την Ευρώπη θα βλάψουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτό ήταν λοιπόν αυτή ήταν ε, η έννοια της ε, συμφωνίας αυτής. Όμως έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα εισαγωγή σόγια, συγκροπημένο φυσικό αερίο, όπως σας ανέφερα και από το σημείο 11, για τη σόγια. Είχαμε και μια ταχύτατη πιστοποίηση των σπόρων σόγιας υπό την οδηγία για την ενέργεια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ρησόγειο για το βιοντίζελ. <coughs> Um, uh, Ελήφθησαν λοιπόν αρκετές δράσεις προς την πλήρωση αυτής της συμφωνίας. Τώρα, σε σχέση με τον ΠΟΕ, μόλις είχαμε αυτό το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά του Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, ο κύριος Σλιμενέκ ε, γνωρίζει αυτή την επιτροπή, είχε εξαφανιστεί όμως και είχε πάει στο Παρίσι, στον ΩΣΑ, αλλά έχει επανέλθει. Και τώρα το καθήκον του είναι να μας εξηγήσει ποια καταπληκτική πρόοδο έχουμε πετύχει μετά την κοινή δήλωση του 2018. Ja, vielen Dank, Herr Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ήρθα να σας ενημερώσω και σας και τα με... της Επιτροπής Ίντα σχετικά με την πρόοδο που έχουμε δει. Μετά τον Ιούλιο άρχισε το πρόγραμμα εργασίας μετά την συμφωνία Juncker-Trump από τον Ιούλιο του 2018. Από τότε δημιουργήθηκε εκτελεστική ομάδα εργασίας για να δούμε τις διάφορες συνεργασίες που θέλαμε. Έχουμε πολλά μικρά θετικά ωφέλη που ως ένα βαθμό εμείωσαν τις εντάσεις θεωρούμε και ενθάρρυναν κάποια συνεργασία όχι τόσο όσο αναφέρατε αλλά κάποιες συνεργασίες ε, διμερώς και συνεργασίες με τις ΙΠΑ επί διαφόρων προκλήσεων. Ορισμένες έχουν ε, γίνει πιο πιεστικές. Ας δούμε πρώτα το διμερές ζήτημα που, της έκθεσης προόδου που είδαμε από τον Ιούλιο που ήταν ένα μεγάλο έγγραφο που εξέταζε ε, τη ροή των εργασιών Κάναμε κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές υγροποιημένου αερίου. Ε, επίσης διαφοροποίησαμε το τομέα της γεωργίας ε, με την εισαγωγή σόγιας. Ε, έγιναν επίσης, έγινε μια οριζόντια συμφωνία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και πολλά, πολλές τεχνικές σημαντικές συζητήσεις περί θεμάτων ρυθμιστικών αν συμφωνήσαμε για την ε, αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη ΣΥΠΑ, οι εξαγωγείς πολλών τομέων θα μπορούν να πιστοποιούν τα προϊόντα τους στη χώρα τους. Θα μπορούμε στην Ευρώπη δηλαδή να πιστοποιούμε εξαγωγές της ΣΥΠΑ και αντίστροφα. Και θα γίνει μια πρόταση σχετικά. Από την άλλη πλευρά ζητήσαμε και κάποιες δεσμεύσεις στο τομέα των μηχανημάτων και πρέπει να δούμε την αντίδραση των ήπα σε όλα αυτά. Σε άλλους ρυθμιστικούς τομείς, τεχνικούς, αλλά ε, σημαντικούς ε, από οικονομικής πλευράς, φάρμακα, ιατρικά μηχανήματα. Έχουμε ενισχύσει ήδη τη συνεργασία μας. Ε, τον Ιούλιο στα φαρμακευτικά προϊόντα ε, καταλήξαμε στις ε, βέλτιστες παρασκευαστικές πρακτικές. Για... Ε, ε, παλιά θα έπρεπε να έρθει επιθεωρητής από την άλλη χώρα για να κρίνει τις εγκαταστάσεις και την παρασκευή των προϊόντων. Τώρα ε, υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, στο, στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης αναγνωρίζουμε τα συστήματα ο ένας του άλλου και αυτό εξικο... μειώνει πολύ το κόστος. Επίσης οι επιθεωρητές που έχουμε εμείς και οι Αμερικανοί μπορούν να πάνε αλλού, σε άλλες χώρες του κόσμου αν θέλετε, για να εξετάσουν την ασφάλεια και τις πρακτικές ε, παραγωγής ε, φαρμάκων. Θα υπάρξει και άλλη πρόοδος, γιατί τα φάρμακα είναι ένα. Τώρα ε, εξετάζομαι και τα κτηνιατρικά φάρμακα, εμβόλια, πλάσμα, που είναι διαφορε... υπάρχουν εκεί διαφορετικοί κανόνες, αλλά είναι πολύ πρακτικά θέματα αυτά που εξοικονομούν πολύ κόστος. Τώρα για τα ιατρικά μηχανήματα δεν θέλω να πλήξετε με τις λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να υπάρχουν βιομηχανίες που να ενδιαφέρονται. Για τα ιατρικά μηχανήματα διευκολύνω με κάποια συστήματα ελέγχου, ε, ένα πρόγραμμα ενιαίου ελέγχου για τα ιατρικά μηχανήματα, που σέβεται για τη δική μας νομοθεσία και διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση αυτών των πρακτικών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κάτι άλλο δύσκολο οι μοναδικοί αναγνωριστές των συσκευών είναι ένα σύστημα που επιβαρύνει πολύ και θα διευκόλυνε να ευθυγραμμίζαμε την ε, το σύστημά μας για να εντοπίζουμε και να ε, αναγνωρίζουμε συσκευές. Επίσης για τα πρότυπα έχουμε κάνει προτάσεις για τα πρότυπα στη ΣΥΠΑ και για τις αναδυόμενες τεχνολογίες ιδιαίτερα. Τα πρότυπα είναι οι, νέες, ε, οι νέοι δασμοί. Άμα με τα πρότυπα έχετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πλέον και ενώ για πολλά χρόνια οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κυριαρχούσαν σε αυτό το τομέα, σε όλο τον κόσμο, τώρα έχουμε την Κίνα που είναι μεγάλος ανταγωνιστής που έχει πολιτική μέχρι το 2025 να αναπτυχθεί πάρα πολύ και αυτό είναι πρόκληση για τους τομείς μας. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τους ΙΠΑ για τα νέα αναδυόμενα πρότυπα, πάρα πολύ περίπλοκα γιατί υπάρχει και διαφορά κουλτούρας που επηρεάζει και τα πρότυπα. Κάναμε προτάσεις όμως, ε, ζητήσαμε προτάσεις από τους εμπλεκομένους, πήραμε 62, είναι στο website και ε, τώρα θέλουμε να γίνουν πιο εύχριστα για να εντοπίσουμε νέους τομείς συνεργασίας με τις ΕΠΑ και ε, σύντομα θα έχουμε νεότερα εδώ. Ξαναγυρίζω στην κοινή δήλωση και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, ε, δηλαδή η ιδέα να αρχίσουν συζητήσεις για την κατάργηση των βιομηχανικών δασμών. Έχουμε διαπραγματευτική εντολή εδώ για να προχωρήσουμε. Και εδώ έχουμε κολλήσει, αν θέλω να είμαι γιατί οι Αμερικανοί έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση και Καταλαβαίνετε ότι η κόκκινη γραμμή για μας είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν να βάλουν μέσα και τους γεωργικούς δασμούς. Αυτό δεν ήταν μέρος της εντολής ούτε της αρχικής ιδέας ούτε ε, ο πρόεδρος της Κομισιόν θα συμφωνούσε. Θα ξεκαθαρίσει τη θέση του και ο νέος πρόεδρος. Θα δούμε λοιπόν εδώ τι πρόοδο μπορούμε να έχουμε. Ε, πάντως ε, γίνονται πολλές εργασίες για την, ε, το θέμα της τρίτης χώρας. Εδώ έχουμε θέματα με τις επιδοτήσεις, ε, αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς, γιατί εδώ οι κρατικές ε, επιχειρήσεις κάνουν εξαγωγές. Επίσης η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας είναι μεγάλο θέμα. Έχουμε θέματα με τη ΣΥΠΑ σε αυτό το τομέα, γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή θα πάνε στον ΠΟΕ. Αλλά έχουμε μια κοινή προσέγγιση ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση ο ΠΟΕ και εργαζόμεθα με τους ε, Αμερικανούς όπου μπορούμε, στους τομείς όπου συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό γίνεται και με τις ΙΠΑ αλλά και με τους Ιάπωνες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα για να με εταίρους για να εξυγχρονίσουμε τον ΠΟΕ. Συνοψίζω, η απερχόμενη Επιτροπή εργάστηκε επί τη βάση της ε, συμφωνίας Juncker-Trump και εσείς το είπατε κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί, να τίνουμε χείρα βοηθείας, να έχουμε θετική ατζέντα με τον ε, εταίρο μας. Η νέα Επιτροπή θα τα ξαναδεί με καινούριο μάτι όλα αυτά, ε, μια φρέσκια ματιά, να δούμε τι πρέπει να ξαναμελετήσουμε, να τροποποιήσουμε κλπ. Να ενημερώσουμε. Είμαστε σε σύνθετη φάση για να το πω έτσι, επίκειται συμφωνία Airbus. Ε, έχω, ε, νομίζω ήρθε πια η απόφαση, έχουμε σαφείς ενδείξεις από εκεί. Επίσης έχουμε και τους Μεξικανούς που θέλουν να απαλλαγούν από τις, τους δασμούς στο Χάλιβα και ε, αντιμετωπίζουμε την απειλή δασμών για την αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε λοιπόν και τις αποκλήσεις που υπάρχουν στον ΠΟΕ, αλλά στον ΠΟΕ και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είναι θετικά τα αποτελέσματα χωρίς να είμαστε και απλοϊκοί. Τώρα, για τα αεροπλάνα, εδώ είναι διαφορετικό το θέμα, γιατί και η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα προσκρούσουν στους, ε, στα νομικά ζητήματα που θέτει ο ΠΟΕ. Ε, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε η μία ή η άλλη πλευρά να επιβάλλουν αντίμετρα με τη μορφή δασμών, αλλά αυτό θα έβλεπτε, θα έβλεπτε και τους δύο. καλό είναι να κατανοήσουμε ότι αυτά τα προβλήματα δεν είναι, τα, μεγάλα προβλήματα δεν είναι μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε σοβαρούς ανταγωνιστές, ε, νέους, νέους εισερχόμενους στην αγορά που μπορεί να μας απειλήσουν. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει συνεργασία γιατί υπάρχουν πολλές νέες κρατικές ε, επιχειρήσεις που μπορεί να είναι ε, αποτελεσματικές. Ε, έχουμε λοιπόν προτάσεις, καταστήσαμε στις σαφές της είπα ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε και το κάναμε αυτό και πριν από το καλοκαίρι με πολλούς τρόπους, αλλά ναι, και μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι οι Αμερικανοί θα αρχίσουν ειλικρινώς διαπραγματεύσεις. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Συγγήτης, μία ερώτηση. Ο λόγος του όλου αυτού εγχειρήματο της κοινή δήλωσης ήταν η δασμή για το χάλιβα και το αλουμίνιο. Συνήθως δεν εστιάζω στους δικούς μου ψηφοφόρους, αλλά υπήρχε μια χαλιβουργία που θύχτηκε από τους δασμούς dumping κατά 22,2% και μετά επιπλέον ήρθε και το 25%. Ε, Συνολικά δηλαδή γύρω στο 50% για τις εξαγωγές χάλιβα που είχαν. Αυτό φυσικά ότι ε, σημαίνει ότι έχει ε, σταματήσει η συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό λίγο πολύ έγινε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και έτσι ε, γι' αυτό έκανε όλη αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποκλιμάκωση κλπ. Μπορείτε να μου πείτε ποια πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί στη συζήτηση για την ε, κατάργηση αυτών των δασμών που δεν ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες του ΠΟΕ. Και υπάρχουν άλλα βήματα που έχουν γίνει ώστε να αρθούν αυτοί οι δασμοί στο χάλιβα. Ειλικρινά, μακάρι να είχα την απάντηση. Το θέτουμε αυτό το ζήτημα σε κάθε ευκαιρία που έχουμε και όσο πιο έντονα μπορούμε και όπως ξέρετε πήραμε και εμείς αντίμετρα που είναι νόμιμα κατά τη γνώμη μας. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα κακό παράδειγμα με ένα άλλο κακό παράδειγμα. Πήραμε τα μέτρα που θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητα και που άξιζε να ληφθούν, πιστεύω. πρέπει να περιμένουμε να ενσωματωθεί η λογική αυτή και η συνειδητοποίηση μέσα στο σύστημα ε, και δεν θέλουμε να κινηθούμε έξω από τους κανόνες του ΠΟΕ. Ναι, είναι σαφές λέει αυτό ο πρόεδρος, αλλά για να συνοψίσω. Εμείς κάναμε πολλά σαφή βήματα προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ και όσον αφορά το χάλιβα και το αλουμίνιο και τις, ε, τους δασμούς δηλαδή που επιβλήθηκαν εκεί, δεν υπάρχει καμία μετακίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, ο κύριος, η κυρία Σράινε Μάκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ανέφερα προηγουμένως, χαίρομαι που ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια επικοδομητική και υπεύθυνη στάση στη, στο θέμα αυτής της συμφωνίας, αλλά πραγματικά ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι έχουν κάνει το δικό τους κομμάτι με τη σόγια, το υγροποιημένο αέριο, τις συμφωνίες για τη συμβατότητα. Αναρωτιέμαι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε πραγματικά τηρούν τις υποσχέσεις τους. Ακούω την Κομισιό να λέει ότι έχουμε κολλήσει ε, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ε, μείωση των ε, δασμών για τα βιομηχανικά αγαθά και αναρωτιέμαι. Ε, βέβαια δεν είναι γεωργικά αυτά τα προϊόντα, αλλά συζητήσαμε μόλις το θέμα της εισαγωγής βοήου κρέατος ε, χωρίς ορμόνες. Θα μπορούσε λιγάκι να βοηθήσει αυτό ε, τις ΗΠΑ να μετακινηθούν στις θέσεις τους. Η κίνησή μας δηλαδή όσον αφορά το βόηο κρέας. Ναι, ευχαριστώ για την παρουσίαση, λέει η επόμενη ομιλήτρια. Ο πρόεδρος Τραμ δεν έχει αλλάξει θέση του τελευταίο καιρό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισαγωγικοί δασμοί για χάλιβα και αλουμίνιο συνεχίζουν να ισχύουν και συνεχίζει να μας απειλεί για επιβολή δασμών για αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μπλοκάρει τον ορισμό ε, δικαστών στον ΠΟΕ. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση στα πλαίσια της προεδρικής αυτής θητείας. Η Κομισιόν ελπίζει ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την περσινή κοινή δήλωση του Ιουλίου ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα και ότι θα, θα παίξουν και οι δύο πλευρές ε, σύμφωνα με, το, με τους κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για την ενημέρωση. Τον κατάλογο των προβλημάτων τον ανέφερε ο πρόεδρος πολύ ωραία. Θα με ενδιέφερε το εξής. Εμείς κάνουμε μονόπλευρα βήματα προς τις ΙΠΑ και ίσως γινόμαστε έμεσα συνεργοί του εμπορικού πολέμου από πλευράς ΙΠΑ προς εναντίον άλλων. Ε, ο χάλιβας, η σόγια που την εισάγει από τη Βραζιλία εντωμεταξύ. Όποτε μπορεί. Όχι, όχι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα, εμείς εισάγουμε αθώα σόγια σε μεγάλες ποσότητες από τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή πρέπει να δούμε και γεωπολιτικά πώς έχει το θέμα και πώς θα διαμορφωθούν οι εμπορικές σχέσεις ε, με τις ΗΠΑ και μέσα με τις άλλες χώρες. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Τρίτον, η Süddeutsche Zeitung γράφει τον Ιούλιο ε, προσοχή, ο Ντόναλτ Τραμπ έχει κάνει το δολάριο όπλο στον εμπορικό πόλεμο. Και αναφέρονται πολλά σενάρια τα οποία παρακολουθεί η Wall Street ε, σε βάρος άλλων ε, νομισμάτων και χωρών. Ερωτώ λοιπόν την Κομισιόν τι συνέχεια θα δοθεί σε όλα αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την εμπορική στρατηγική που ίσως θα τεθεί και από το νέο Επίτροπο υπεύθυνο για το εμπόριο ε, που θα αναφερθεί στις δικές μας προσδοκίες, αλλά στον διμερή διάλογο, όταν γίνεται αναφορά σε κοινούς στόχους και αξίες κλπ, θα πρέπει να δοθεί απάντηση στις καινούριες αυτές ε, ε, εμπορικές πρακτικές που δεν, δεν, δεν προάγουν τα συμφέροντά μας αλλά και το διεθνές εμπόριο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα, τι θα κάνουμε, ε, θα κάνουμε χωριστές συμφωνίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα ή τα γενώσιμα ε, που προωθούν οι Αμερικανοί στις άλλες αγορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εμπορική συνεργασία κατακαιρματίζεται τρόποντινά ε, και έτσι χάνουμε τον γενικότερο στόχο από τα μάτια μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσει η Κομισιόν μια ανοιχτή επιστολή που στάλθηκε από πολλές ε, ΜΚΟ στην ε, κυρία Ούρσουλα Φοντελέιεν ε, και στον κύριο Χόγκαν σε σχέση με το θέμα της διαφάνειας και ε, τονίζουν οι ΜΚΟ για τις διαπραγματεύσεις ότι αντίθετα με όσα συμφωνήθηκαν οι διαπραγματεύσεις ε, δεν αφορούν ένα περιορισμένο αριθμό ζητημάτων αλλά και ότι δεν είναι και τόσο ανοιχτέ ούτε διαφανείς. Διαβάζοντας την έκθεση της σύνοψης κατόπιν της διαβούλευσης ε, τον Ιούλιο ανησυχώ με τον ενθουσιασμό που δείχνει η Κομισιόν απροκάλυπτα για την συμμετοχή των επιχειρήσεων και το ότι οι τομεί τη συνεργασία είναι ευρύτεροι από αυτού που αρχικά είχαν τεθεί. Έτσι λοιπόν, ε, μήπως ε, θα δημοσιεύσετε τα έγγραφα και θα αποκλείσετε τους τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην εντολή του Συμβουλίου. Και επίσης δεσμεύεστε να κάνετε και μελέτες αντικτύπου στο επίπεδο των δικών μας προτάσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάντη. Πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Αν εγώ έπρεπε να ορίσω τον τόνο αυτής της συζήτησης, ε, το ύφος της, ε, θα έλεγα ε, το ε, σύνθημα ότι εδώ έχουμε απλά και μόνο να ελπίζουμε. Δηλαδή, βρισκόμαστε στην κατάλληλη στιγμή όπου ε, καταδικάζει την Ευρώπη και δίνει τη δυνατότητα στον Τραμπ να βάλει δεσμού 12 δισεκατομμυρίων και αυτοί θα πέσουν όχι στην ευρωπαϊκή αεροπλοεία αλλά στους γεωργούς 4 δισεκατομμύρια ε, θα αφορούν την Ιταλική ε, τον Ιταλικό γεωργικό κλάδο και μάλιστα διαβάσαμε και το Twitter της Επιτρόπου Μάλστρομ που είναι η αρμόδια επίτροπος αυτή τη στιγμή. Συζητάμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά φαίνεται ότι σήμερα είμαστε εκτός πλαισίου. Δεν είμαστε σε μια στιγμή στην οποία θα πρέπει φυσικά να ενισχύσουμε την ελπίδα απέναντι σε αυτή τη συμφωνία ξέρουμε ότι πάντοτε οι δασμοί είναι κάτι κακό και φυσικά πλήττουν την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά πλήττουν και την αμερικανική οικονομία. Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι δύσκολο να το δούμε αυτό σε ένα μήνυμα ελπίδας αυτή τη στιγμή σε σχέση με το τι βιώνουμε. Έτσι λοιπόν, ρωτώ, ποιον αντίκτυπο θα έχει η τελευταία απόφαση σε διαπραγματεύσεις που φαίνεται σήμερα να είναι εκτός ιστορίας και εκτός ε, πλαισίου. Um, Κοιτάξτε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Yes, thank you, I have to... Ναι, ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι ανησυχώ γιατί ο Τραμπ μας αναγκάνει να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνσή του σιγά σιγά, βηματάκι βηματάκι. Και τελικά πού βρισκόμαστε. Από ό,τι φαίνεται είναι σαν να γδινόμαστε μπροστά στον Ντόναλτ Τραμπ και τελικά θα μείνουμε εντελώ γυμνοί πρέπει να σκεφτούμε ποια θέση θα λάβουμε. Και για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Ντάντη. Εγώ διάβασα 7,5 δισεκατομμύρια, είπατε 12 δισεκατομμύρια σε δασμούς, αλλά είχατε δίκιο στο εξή ότι πολλά γεωργικά προϊόντα θα είναι στον κατάλογο του Ντόναλτ Τραμπ. Και αυτή είναι μια ερώτηση που έχει ήδη τεθεί σε διάφορες συναντήσεις βλέπω ότι ο Ντόναλτ Τραμπ προσπαθεί να εφαρμόσει το διέρη και βασίλευε, γιατί τα ιταλικά προϊόντα, τα γαλλικά προϊόντα θα είναι αυτά που εκτίθενται περισσότερο στον κατάλογο αυτό και θα προσπαθήσει να σπάσει την ενότητα των κρατών μελών για να πούν άλλοι ότι είμαστε τελικά δεν μας ενδιαφέρει. Αν και αυτό δεν ισχύει, πώς θα εγγυηθεί η Κομισιόν ότι θα διατηρηθεί η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί ο Τραμπ προσπαθεί εδώ να μας διασπάσει. Ξέρετε, όταν έρχεται ο λύκος, αρχίζουν τα πρόβατα να τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Και θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Τιτσιάνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω εκπλαγεί. Πιστεύω ότι η κοινή δήλωση του 2018 θα χρησιμεύεται για να ξευμενήσει τα πνεύματα, όμως από ό,τι φαίνεται είμαστε ε, μπροστά σε έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ε, και το είχε πει η Κομισιόν ε, τότε, δεχτήκαμε περισσότερη σόγια, και βιοκαύσιμα. Όμως δυστυχώς τελικά στρέψαμε και το άλλο μάγουλο. Τώρα εδώ θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι αυτό αποτελεί κάθετη επίθεση στην ενότητά μας ε, και το γεγονό ότι στοχεύονται συνήθως ε, τα γεωργικά προϊόντα που αφορά αυτό κυρίως στη χώρα μου αποτελεί ε, ουσιαστικά προσπάθεια να διασπαστεί το ευρωπαϊκό μέτωπο και ε, νομίζω ότι ε, το να, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία συμφωνία, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, εγώ είμαι αποφασισμένη να απαντήσουμε με το ίδιο νόμισμα και να δούμε ποια απόφαση μας επιτρέπει ε, να επιβάλλουμε δασμούς 4 δισεκατομμυρίων, αυτό αμέσως ε, θα μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το δούμε. Και να το θέσουμε επιτάπητος. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, για να επανέλθω στα ευρωπαϊκά, είναι ότι κυρίως οι χώρες του Νότου θα πληγούν. Εγώ νομίζω ότι για να αποφύγουμε αυτό το κατακαιρματισμό πρέπει να προβλέψουμε ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης κυρίως για τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Ισπανούς γεωργούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την έκτακτη κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να χρηματοδοτείται από όλους διαφορετικά. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε ε, για διάσπαση του Ευρωπαϊκού Μετώπου όταν η κάθε χώρα θα προσπαθήσει διμερώς να διαπραγματευτεί ε, κρυφές εξαιρέσεις. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο κυνηγός, ποιος θα είναι ε, ο επικεφαλής των λύκων που κυνηγάει τα πρόβατα. Ε, ε, κοιτάξτε, είναι σαν να είμαστε στο ε, ποδόσφαιρο ε, και κάποιος παίζει με κανόνες handball και δεν υπάρχει διαιτητής. Εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε με τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Το πρώτο που κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε τα συμφωνηθέντα του Ιουλίου και αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ε, πρόσχημα να πούν ότι απέτυχε. Άλλωστε υπάρχουν πρόοδοι σε ρυθμιστικά θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας. Μπορεί να μην ανταποκρίνονται αυτά στις προσδοκίες που είχαμε, αλλά κάποια πράγματα γίνανε. Και βέβαια η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού, το ξέρετε αυτό. Προσπαθούμε να πείσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι είναι καλύτερο να συνεργαστούν μαζί μας διμερώς ε, ε από το να επιλέξουν τη μονοπλευρή προσέγγιση. Εμείς πήγαμε στο δικαστήριο, συζητήσαμε, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η επίπτωση όλων αυτών και πολλές φορές ε, υπάρχει ε, επιζήμια επίπτωση όχι μόνο για μας αλλά και για εκείνους, Αυτά, ε, αυτή είναι η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Και να μπορούμε να συζητήσουμε και να προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, και να δούμε κάποιους κανόνες που θέτουν η Κίνα και άλλες ισχυρές αναπτυσσόμενες χώρες ε, καλύτερα να μην κλιμακώσουμε ε, την ένταση ε, με ένα σημαντικό εταίρο. Δεν χρειάζεται να σας δείξω με νούμερα πόσο σημαντικοί εταίροι είμαστε. Είναι αντιπαραγωγικό να μην συνεργαζόμαστε. Και εξετάζοντας τη συμφωνία μπορώ να πω ότι έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα, σύντο χρόνο θα κάνουμε και άλλες πρόοδους. Είναι σαφές ότι αυτό που κάνουμε και το είπατε κάποιοι, μιλήσατε και για τη διαφάνεια, η διαφάνεια είναι σημαντική. Ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες. Υπάρχει βέβαια δημόσια κριτική, αλλά εμείς προσπαθούμε να κινηθούμε στα πλαίσια της εντολής μας. Αυτό είναι σαφές αλλά εξίσου σαφές είναι ότι αν υπάρχει ε, διαφορετική τροπή στις ε, διαπραγματεύσεις θα γίνει μελέτη επιπτώσεων και ελπίζω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα πιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι πρόκειται για μια μοναφίντε ε, προσπάθεια. Τώρα για το Airbus και τη σημασία του καλό θα ήταν να ξεχωρίζουμε τα θέματα. Η Airbus και η Boeing, που κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε και αυτό, είναι νομικές διαδικασίες. Ατυχές με ένα, καλά να ακολουθείτε τους κανόνες, αυτή είναι μια συνέπεια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, κάνουμε συνδέσεις με τα άλλα διμέρη θέματα που κατά τη γνώμη μας είναι παράνομα. Ε, θα πρέπει να πούμε στους Αμερικανούς, αυτό που είπε και η κυρία Μπέγκιν, ότι αν θέλουν πόλεμο ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να αποκριθούμε έτσι και θα αξιοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε, δεν θα καθίσουμε να τις τρώμε. Θα πρέπει να δούμε πάντως πρώτα τι πρόοδος θα υπάρξει ε, στη, στα αεροπλάνα και στα ανταλλακτικά τους. Θα δούμε. Και ε, πρόσκληση για ενότητα ε, ε, υπάρχει. Μπορεί να είμαστε μαζί, θα δούμε βέβαια ε, τι πολιτική συνεννόηση μπορεί να υπάρξει. αν ισχύουν ίσοι οι κανόνες του παιχνιδιού, που ελπίζουμε ότι θα ισχύσουν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τον οριστικό κατάλογο και μετά θα δούμε τι πρέπει να γίνει και να ε, ξεκαθαρίσουμε στις ΕΙΠΑ ότι ε, αν κινηθούν προς αντίθετη κατεύθυνση και εμείς δεν θα διστάσουμε μετά από λίγο, λίγους μήνες να κάνουμε αυτά που πρέπει. Αυτά. Αν ξέχασα κάτι, πείτε το μου. Ε, ακούστηκαν πολλά ωραία πράγματα. Πάντως στο βασικό είναι συνεχίζουμε τις προσπάθειες και βέβαια εκτιμούμε την υποστήριξή σας γιατί και εσείς έχετε τον ίδιο προβληματισμό όπως η Επιτροπή. Βέβαια οι Αμερικανοί δεν είναι μονολήθικοι στην, στην κυβέρνηση, υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις. Και εμεί θα πρέπει να έχουμε ενότητα, ε, όχι μόνο η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, αλλά και οι εμπλεκόμενοι για να αντιμετωπίσουν το θέμα. Ο κύριος Κέλλη. Καταρχήν, ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ ε, έκανε μια προσπάθεια να ηρεμήσει την κατάσταση με τη ΣΥΠΑ. Ε, το αποτέλεσμα ήταν η συμφωνία που εφαρμόζουμε. Αλλά σχετικά με την τωρινή απόφαση για το Airbus, από ό,τι κατάλαβα, επιτρέπει στη ΣΥΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις σε εμάς πολύ σύντομα. Αλλά εμείς πρέπει να περιμένουμε μέχρι την απόφαση ε, για τον Boeing την Άνοιξη. Μπορούμε μπορούν να μας καθυστερήσουν, να μην πάρουμε αντίμετρα εμείς και εκείνοι θα έχουν το προβάδισμα έχοντας λάβει μέτρα για 5-6 μήνες. Αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και τις εκλογές τους ο ΠΟΕ μας περιορίζει, μας βάζει σε μειονεκτική θέση, ενώ βάζει εκείνου σε προνομιακή θέση. Ευχαριστώ. Ε, ε το ερώτημα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις διαδικασίες. Γιατί πριν από 15-18 χρόνια πριν αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε τη δική μας την υπόθεση. Δεν αλλάζει αυτό εύκολα. Τι μπορεί να γίνει, να ξεκαθαρίσουμε ότι το σενάριο αυτό που ακούσαμε είναι ένα σενάριο που το έχουμε υπόψη μας και δεν πρόκειται να κάνουμε διαπραγματεύσεις με το όπλο στον κρόταφο, γιατί μέχρι τον Οκτώβριο ελπίζουμε ότι θα έχουμε λύση. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα νομίζω προς εκείνους ότι ο παράγων χρόνος δεν θα λειτουργήσει υπέρ αυτών. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τι να κάνετε, είναι υποχρέωση αυτή ενός μέλους της διοίκησης. Λοιπόν, τελειώσαμε και το σημείο 12 και πάμε στο σημείο 13. Η Ορδανία και μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς αυτήν. Ε, η Ορδανία λοιπόν θα πάρει μακροοικονομική χρηματοδοτική 80 εκατομμύρια το 16 200 εκατομμύρια εγκρίθηκαν και τώρα συζητάμε 500 εκατομμύρια για να δώσουμε στην Ιορδανία. Έχει ήδη λάβει αυτά τα ποσά που σας είπα. Πολλά λεφτά. Και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Σαντιάγκο Λοάνκα Γκαρσία, ε, κεφαλής ε, από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ να παρουσιάσει την πρόταση. Μέχρι πέντε λεπτά χρόνο έχετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, όπως ξέρετε η Κομισιόν στις 6 Σεπτεμβρίου υιοθέτησε μια πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής ε, συνδρομής για το Χασεμετικό Βασίλειο της Ιορδανίας μετά από ένα αίτημα εκ μέρους των Ιορδανικών Αρχών που ε, υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2018. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων, ε, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Ιορδανίας και τους εξωτερικούς παράγοντες, παράγοντες ευαλωτότητας της χώρας και τις οικονομικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος μιας ε, διεθνούς προσπάθειας και με το πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να συμβάλλει στην ε, οικονομική σταθεροποίηση της Ιορδανίας με μακροχρόνια χρηματοδότηση, με ελκυστικούς όρους που θα βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την εφορία του χρέους της και να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που ε, χρειάζονται για την ευημερία της ε, χώρας και για να αντέξει η οικονομία της στις εξωτερικές ε, ε, πιέσεις. Επίσης, αυτή είναι μια υποστήριξη προς μια χώρα που συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια, ειρήνη και ανάπτυξη της περιοχής της και αυτό συμπεριλαμβάνει και την φιλοξενία μεγάλου αριθμού πληθυσμών Συρίων, κυρίως προσφύγων στην Ιορδανία. Η οικονομία της Ιορδανίας συνεχίζει να επηρεάζεται από τις ε, περιφερειακές αβεβαιότητες και ιδιαίτερα από τον αντίκτυπο της ε, σύραξης στη Συρία, ε, με, διότι διάφορες εμπορικές, διάφορες εμπορικές οδοί έχουν μπλοκαριστεί και υπάρχει ε, όπως είπα και σημαντικός αριθμός σύρων προσφύγων. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιους από τους βασικούς δείκτες που παρουσιάζουν τη μεγάλη πρόκληση που αποτελεί η κατάσταση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι μόνο 1,9% ήταν το 2018 και παρόμοιες επιδόσεις αναμένονται και για φέτος, γύρω στο 2% που είναι η χαμηλότερη επίδοση από το 1996. Μετά, η αναγκή για δημοσιονομική εξυγίανση ε, συνεχίζει να υπάρχει παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τις αρχές και η επιτυχία στην μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ε, έχει ε, εν μέρη αντιστραφεί. Ήδη διευρύθηκε το χρέος το 2018 και βλέπουμε περαιτέρω αύξηση του 2019. Κυρίως αυτό οφείλεται σε ε, δημοσιονομικά έσοδα χαμηλότερα από το αναμενόμενο το δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλό επίπεδο, 94% του ΑΕΠ και το μισό περίπου από αυτό το χρέος είναι εξωτερικό χρέος σε δολάρια Αμερικής. Το εμπορικό έλλειμμα παραμένει υψηλό, ε, το έλλειμμα συγγνώμη, παραμένει υψηλό, 7% ε, του ΑΕΠ Υπάρχουν όμως ενθαρρυντικές ενδείξεις όσον αφορά ε, τον δίκτυο αυτό. Ιδίως ε, αυτό οφείλεται σε ε, αυξήσεις των εξαγωγών. Όμως οι άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στο παρελθόν. Τα χρόνια 2005 με 2010 ήταν 12,7% του ΑΕΠ έπεσε στο 4,5 τα χρόνια 2011 έως 2018 και ε, πέρυσι παρέμεινε στο 2,2% του ΑΕΠ. Και τέλος, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των αριθμητικών δικτών, η ε, ανεργία συνέχισε να αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι κάπου πάνω από το 19%, πλήττοντας κυρίως το, τους νέους και τις γυναίκες. Σε αυτό το πλαίσιο η, η πρωτοβουλία του Λονδίνου του Φεβρουαρίου φέτος αποσκοπεί στο να ε, συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας μεταξύ των των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υποστήριξη της ε, Ιορδανίας με μακροοικονομική βοήθεια από δωρητές για να καλύψει η χώρα τις εξωτερικές ανάγκες, να εξυπηρετήσει το χρέος της, την αηφορία του χρέους, αλλά επίσης και για να υποστηρίξει ε, διάφορες μεταρρυθμίσεις ε, για την ανάπτυξη και για ε, τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. Στη διάσκεψη εδώ του Λονδίνου, η Κομισιόν εξέφρασε την ετοιμότητά τη να ε, εξετάσει το ενδεχόμενο ενό τρίτου προγράμματο μακροοικονομική βοήθεια με 200 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δέσμευση ήταν κάτι που επαναλάβαμε πέρυσι την Άνοιξη στη διάσκεψη των Βρυξελών, όπου αφορούσε το μέλλον της Συρίας και της περιοχής. Το ποσό αυτό τελικά, είπε η Κομισιόν, θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση των οικονομικών αναγκών της Ιορδανίας όταν θα έρθει η στιγμή για να κάνει την πρότασή της η Κομισιόν. Λίγους μήνες Αργότερα, το Μάιο του 2019, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ολοκλήρωσε τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης της Ιορδανίας και εκτίμησε το IMF ότι οι οικονομικές ανάγκες της Ιορδανίας είναι 6,4 ε, δισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2021. Ε, Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές της Ιορδανίας φέτος τον Ιούλιο ζήτησαν 500 εκατομμύρια ευρώ ε, επιπλέον μακροοικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να, υποστηριχθούν οι ανάγκες του ισοζυγίου της χώρας και οι ε, υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό. Μετά από μια σε βάθος αξιολόγηση που έγινε ε, της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης της Ιορδανίας, στις 6 Δεκεμβρίου η Κομισιόν υιοθέτησε μια πρόταση για ένα τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι το τρίτο τέτοιο πρόγραμμα και θα ακολουθήσει, ακολουθεί μια δεύτερη ένα δεύτερο τέτοιο πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε πλήρως ε, τον ε, Ιούλιο του 2019 200 ε, εκατομμύριων δολαρίων και το προηγούμενο το πρώτο που ήταν 180 εκατομμύριων δολαρίων. Επίσης η Κομισιόν συνεπής με μια προηγούμενη δέσμευσή της που εκφράστηκε στην απόφαση για τη δεύτερη μακροοικονομική βοήθεια τον Δεκέμβριο του 2016. Οπότε ε, δεσμεύτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν σχετικά με τις απαιτήσει που θα ίσχυαν και ότι αν ίσχυαν οι προϋποθέσεις ε, δεσμεύτηκαν τα τρία όργανα ότι η Κομισιόν θα υπέβαλε ένα τρίτο πρόγραμμα ε, ε, μακροοικονομικής βοήθειας μεγαλύτερου ποσού αν το δικαιολογούσαν οι συνθήκες. Προτείνουμε λοιπόν αυτό το ποσό το οποίο αναμένουμε να καλύψει γύρω στο 10% των οικονομικών αναγκών ε, της χώρας για την περίοδο 2020-2021. Το ποσοστό αυτό λαμβάνει ήδη υπόψη την υποστήριξη από το IMF και την Παγκόσμια Τράπεζα. Το ποσοστό αυτό πιστεύουμε ότι είναι αρκετά λογικό, είναι χαμηλότερο από το ποσοστό με το οποίο υποστηρίζουμε την Τινησία, όπου το ποσοστό αντίστοιχα είναι 20% ή την Ουκρανία. Θεωρούμε όμως ότι ε, είμαστε στο σωστό σημείο ισορροπίας. Το κενό που υπάρχει ε, το, το υπόλοιπο ε, αναμένουμε να καλυφθεί από το Δούνου και την Παγκόσμια Τράπεζα και από τη διεθνή κοινότητα σε διμερείς και πολυμερείς δωρές, μεταξύ των οποίων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και 1 δισεκατομμύριο περίπου θα καλυφθεί με έκδοση ευρωομολόγων στην ε, ιδιωτική χρηματοοικονομική αγορά. Παρόλες όλες αυτές τις βοήθειες παραμένει ένα κενό, 1,7 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια όλων αυτών των θεσμών θα καλυφθεί. Προβλέπονται τρεις δόσεις που εξαρτώνται από μία σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα περιληφθούν σε ένα μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί ανάμεσα στην Κομισιόν και την ε, χώρα. Επίσης ε, εξαρτώνται οι δόσεις αυτές από το πρόγραμμα του Δουνουτού γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα του Δουνουτού το οποίο λύγει του χρόνου το Μάρτιο και αυτοί ήδη έχουν αρχίσει και οι δύο πλευρές να διαπραγματεύονται ε, ένα νέο πρόγραμμα. Και Βεβαίως ε, υπάρχουν και όροι που αφορούν τις πολιτικές συνθήκες, ε, σεβασμό στη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, ε, κράτο δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα. Η απόφαση για τη χορήγηση της βοήθειας αυτής εξαρτάται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μετά από τις συμφωνίες του παρελθόντος, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε το ίδιο μοντέλο για την πρόταση αυτή. Μόνο μια τεχνική τροποποίηση γίνει στο άρθρο 6 και αυτό οφείλεται στις αλλαγές που έγιναν στο δημοσιονομικό κανονισμό του 2018. Ε, άλλαξε ο κανονισμός και πήραμε ακριβώς τη διατύπωση που υπάρχει στον ε, ε, δημοσιονομικό κανονισμό συμμορφούμενη πλήρως. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία ανάμεσα σας, εμάς και το Συμβούλιο, ώστε η πρόταση αυτή να εγκριθεί το γρηγορότερο δυνατό και να εφαρμοστεί, ελπίζουμε, και μέσα στο 2019. Ευχαριστούμε. Να καλέσω τώρα τον κύριο Ντανιέλ Αρίστη, ο οποίος ε, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος για τη Μέση Ανατολή της Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης. Να μας δώσει και τη δική του οπτική για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι αρκετά σύντομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ορδανία έχουν εξαιρετικέ σχέσει. Βασίζονται σε συμφωνία σύνδεση και τις προτεραιότητε ε, της εταιρική σχέση ε, που συμπεριλαμβάνονται εκεί και θεωρούμε ότι οι χώρες μας ε, είναι σύμμαχοι σε μια δύσκολη περιοχή η ίδια η Ιορδανία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, υπάρχει περιφερειακή αβεβαιότητα και ήδη αναφέρθηκε και ο, ρυθμός, ο μεγάλος αριθμός προσφύγων στη χώρα. Ε, υπάρχουν μια σειρά οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων και υποστηρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα στην Ιορδανία και κατά συνέπεια σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν που βρίσκονται σήμερα εδώ για μένα. Είναι μεγάλη τιμή που διορίστηκε εισηγήτρια για την ε, ομάδα του, τον χώρο του Μασρέκ. Σήμερα συζητάμε την ε, πιθανή χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ε, στο βασίλειο της Ιορδανίας, το οποίο έχει πληγεί η σειρά από τη δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση στις όμορες χώρες, στη Συρία και στο Ιράκ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε μια φίλη χώρα όπως η Ιορδανία που αυτά τα χρόνια έχει ε, δει ε, ε, να, τον αντίκτυπο ενός εκατομμυρίου 300.000 προσφύγων από τη Συρία. Έχει υπάρξει και μείωση του τουριστικών ροών και μείωση και του φυσικού αερίου. Χρειάζεται λοιπόν διεθνή και ευρωπαϊκή βοήθεια η Ορδανία για να μπορέσει να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, για να συνεισφέρουμε στη σταθεροποίηση της περιοχής και για να υπάρξει έλεγχος των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ευρώπη δεν μπορεί παρά να υποστηρίξει την Ιορδανία στις προσπαθίες της τα τελευταία χρόνια που έχουν καταστεί δυνατές και ε, χάρη δανείων από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και χάρη των χρηματοδικών συνδρομών. Το 2013 είχαμε 180 εκατομμύρια ευρώ, το 2016 200 εκατομμύρια ευρώ ε, και ε, ουσιαστικά πληρώνονται στι προθεσμίες που έχουν προβλεφτεί. Τώρα μα ζητά νέα οικονομική βοήθεια η Ορδανία 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τρει δόσεις προκειμένου να εξηγιάνει τα οικονομικά τη Σημαντική στήριξη για μια χώρα που καθημερινά καταπολεμά την Ισλαμική τρομοκρατία και είναι κεντρικός ο ρόλος της στη σταθεροποίηση της περιοχής. Επίσης, ε, στο Φεβρουάριο του 2019, στη διάσκεψη του Λονδίνου, οι διεθνείς και περιφερειακές δωρητόες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, επανέλαβαν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν οικονομικά τις προσπάθειες της Ιορδανίας, βοηθώντας την αδιατήρηση μακροοικονομική σταθερότητα και βοηθώντα τη στην ανάπτυξη. Είναι για μα θεμελιώδε η Ορδανία να συνεχίσει τη, διάδρο... τη διαδρομή τη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων ε, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομία τη και να προβεί σε διαφορετικέ μεταρρυθμίσει ε, υπέρ των πολιτών. Επίσης, η χορήγηση της μακροοικονομικής συνδρομής ε, ορίζεται από την παροχή κάποιων εγγύσεων από την Ιορδανία, δηλαδή την απέτηση να διατηρηθούν δημοκρατικοί μηχανισμοί, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη είχαμε θετικά μηνύματα το 2018 ε, με την επανέναρξη της εισαγωγής του αερίου και την άνοδο του τουρισμού. Όμως υπάρχουν ενισχυτικά στοιχεία για την ανεργία, τον πληθωρισμό και για το βαρύ δημόσιο χρέος. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει εγγυητής για το πώς ε, θα δοθούν αυτά τα κονδύλια τα επόμενα χρόνια και ε, να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης είναι θεμελιώδες ε, να δοθούν αυτή, να δοθεί αυτή η οικονομική βοήθεια για την εξισορρόπηση του ισοζυγίου προκειμένου να μειωθεί το αντίκτυπο, ο αντίκτυπος της κρίσης των προσφύγων. Ε, θα ήθελα να προχωρήσουμε με αυτό το σημαντικό φάκελο για το όφελο όχι μόνο της Ιορδανίας που θέλει να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα αλλά και για το όφελος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. κυρία Μπρικμού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας διάβασα στον γράφο εργασίας του προσωπικού στις 6 Σεπτεμβρίου ότι για να ε, λάβουν μακροοικονομική συνδρομή, οι χώρε θα πρέπει να σέβονται το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές αρχέ και να εγγυώνται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ισχύει ότι οι πολιτικές προποθέσει πληρούνται. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ωστόσο, διάβασα κάποιε γραμμές παρακάτω ότι υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, υπάρχουν βασανιστήρια ε, και ελευθερία της έκφρασης και του συνεστερίζεστε. Είναι πολύ δύσκολη η περιφερειακή κατάσταση και το πλαίσιο, όμως δεν μπορούν να αιτιολογηθούν όλα αυτά έτσι λοιπόν αναρωτιέμαι ε, για το αν οι προϋποθέσεις που συνοδεύουν τη χρηματοδοτική συνδρομή ε, πράγματι ε, διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρόοδος και διαφορετικά αν βάσει του άρθρου 212 που παραπέμπει και στο άρθρο 21 δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ε, μακροοικονομική συνδρομή ως μοχλό για να έχουμε σημαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο αυτό. Επίσης, έχω και μια ακόμη ερώτηση. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τη συνδρομή με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας με τις χώρες του Νότου. Εξάλλου, τα 500 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα δάνειο που θα επιστραφεί και αν ναι με ποιο επιτόκιο και με ποια λήξη ή ε, πρόκειται ουσιαστικά για ένα κονδύλι διεθνούς ελληνικής που δίνουμε σε μια χώρα που δέχεται πρόσφυγες και είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα. Τι σημαίνει ότι τα προηγούμενα δύο δεν πετύχαν τους στόχους. Ποιοι ήταν οι λόγοι της αποτυχίας και ποια διδάγματα αντλήθησαν από την ε, αξιολόγηση αυτού του προγράμματος και βάσει κάποιων ε, πρόσφατων δεδομένων η ορδενία με το Ισραήλ ε, μαζί με το Ισραήλ και τη Συρία ήταν η χώρα που είχε πληγεί περισσότερο από τις ανισότητες και ήταν αυτός ε, λόγος για την φυγή ενός εκατομμυρίου προσφύγων. Υπάρχουν πράγματα που προβλέπονται με ακρίβεια για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τις ανισότητες. Ε, καθώς ε, η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι θέλει και να τη θασεύσει την παγκοσμιοποίηση και μας το είπε και ο κ. Χόγκαν τη Δευτέρα και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Κομισιόν ε, σκοπεύει να το συζητήσει αυτό το θέμα και να το συμπεριλάβει στο μνημόνιο συνεννόησης. Επίσης, η συνδρομή θέλει να προωθήσει διευθυντικές μεταρρυθμίσεις για την μείωση της ενεργείας και να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κάλσπρου. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρου του κυρίου Τζέρεμι Ντισάιερ, που ζητά συγγνώμη που δεν παρευρίσκεται εδώ σήμερα το απόγευμα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Εκ μέρου τη ομάδα Ρινιού, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή τη και θέλω να εκφράσω τις ανησυχίες μας σε σχέση με τις δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζει η Ερδονία λόγω της περιφερειακής αστάθειας. Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή, να μεταρρυθμιστεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις σταθερότητε σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Η ομάδα μας λοιπόν θα μπορέσει να υποστηρίξει την ε, υιοθέτηση αυτού του τύματος για μακροοικονομική συνδρομή. Όμως, όπως στο παρελθόν έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της ε, προηγούμενου αιτήματος ε, χρηματοοικονομικής συνδρομής θα δώσουμε προσοχή στο να πληρούνται τα ευρωπαϊκά κριτήρια που συνδέονται με την χορήγηση αυτής της συνδρομής. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, αυτά είναι καθήκον του Κοινοβουλίου, όντως. Ο κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Απλώ να πω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το τελικό κείμενο συνάδει απόλυτα με την πρόσφατη χρηματοοικονομική συνδρομή που θετήθηκε για άλλε χώρες και ε, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επικαιροποίηση και κατάλληλη εφαρμογή σύμφωνα με τους σκοπούς. Ευχαριστώ. Τέλεια. Για να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Μάλλον ε, είναι πολλές οι προκλήσεις που μου θέσατε. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν αρκετά πλήρης οι ερωτήση σας. Όπως είπε και η συγγήτρια. Αυτή η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ε, έχει, συνοδεύεται και από κάποιες προϋποθέσεις. Ανέφερα ότι έχουμε τρεις, τρία είδη προϋποθέσεων. Καταρχήν πολιτικές προϋποθέσεις, και ήδη εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες για το αν η χώρα πράγματι σέβεται αυτές τις πολιτικές προϋποθέσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει εδώ να είμαστε κάπως ευέλικτοι. Δηλαδή να βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα και την τάση για το αν έχουν υπάρξει βελτιώσεις ή όχι στην κατάσταση. Και η άποψη της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι θετική. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και αυτό αποτελεί μέρος της απόφασης. Κάθε εκταμίευση θα είναι υπό προϋποθέσεις για το αν θα συνεχίσουν να σέβονται το δημοκρατικό μηχανισμό, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, οποιαδήποτε επιδείνωση μπορεί να διακινδυνεύσει την εκταμίευση της βοήθειας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι για το ποιες μεταρρυθμίσεις μπορούν να υποστηριχθούν με αυτό το μέσο. Η στήριξη αφορά την χρηματοοικονομική σταθερότητα και επίσης θέτει και τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις ε, τυπικά είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης και σχετίζονται με τα οικονομικά συστήματα, με την, ε, τα συστήματα φορολόγησης, με την δημοσιονομική διαχείριση, με τρόπους ε, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών, αλλά και με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό, το επιχειρηματικό περιβάλλον ή θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας και νομίζω ότι ορθώς αναφέρθηκαν και οι ανησυχίε για τις ανισότητες. Ε, βελτιώνουν και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Στον προηγούμενη μακροοικονομική συνδρομή είχαμε τέτοιες προϋποθέσεις για την αγορά εργασίας και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για τα μελλοντικά μεμοράντα. Ήδη είχαμε την εμπειρία με δύο συνδρομές και οι δύο είχαν αξιολογηθεί εξωτερικά και είχαν λάβει θετικά σχόλια από τους εξωτερικούς αξιολογητές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ως καλοί αξιολογητές ε, τι θα σημαίνει και η έλλειψη υποστήριξης γιατί αυτή η υποστήριξη είναι μέρος ευρύτερης διεθνούς προσπάθειας και η συνολική αξιολόγηση θα έλεγα ότι είναι γενικά θετική. Όλη η υποστήριξη και η μικροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έχει συμβάλει στην αποφυγή της επιδείνωσης και στο να διατηρηθεί η Ιορδανία ως ένα σημαντικό σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδος της στήριξης που θα δοθεί θα είναι δάνειο. Εξήγησα πριν λίγε εβδομάδες πώς ε, γενικά λειτουργεί η μικροοικονομική συνδρομή. Αλλά για να καταλάβετε, ουσιαστικά ε, καλούμε αυτό ε, μία πράξη δανεισμού. Πάει η Κομισιόν στις αγορές, παίρνει κάποιο ε, χρέος και ταυτόχρονα με το ίδιο επιτόκιο δανείζουμε τις χώρες. Δεν υπάρχει κάποιο τέλος ε, το οποίο χρεώνουμε στις χώρες. Δηλαδή είναι πολύ καλές οι, αγορές, οι συνθήκες της αγοράς. Ε, ουσιαστικά είναι ε, η καλύτερη λύση που υπάρχει παγκοσμίω. Οι τελευταίες πράξεις φέτος για την υποστήριξη της Τινησίας και της Ιορδανίας ήταν στο 0,5% με μια ημερομηνία λήξης περίπου 17 έτη. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι βοηθά αυτό πάρα πολύ προκειμένου να έχουμε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα τέτοιων οικονομίων όπως της Ιορδανίας. Όλες οι εκταμιεύσεις όπως είπα θα εξαρτώνται από το αν θα υλοποιούνται οι προποθέσει, οικονομικέ μεταρρυθμίσει, παρουσία προγράμματο Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και σεβασμού των πολιτικών προϋποθέσεων. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο, ευχαρίστως. Μισό τα εκατό. Καλό ποσοστό. Ε, επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Στο κείμενο μας αναφέρεται η θετική διάσταση νομίζω ότι η κατάσταση ε, ότι το μέτρο, τα μέτρα που λαμβάνουμε αντιρροπούν την κατάσταση. Θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν υπήρχε η συνδρομή μας. Ευχαριστώ. Σίγουρα σταθεροποιείται η κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πρόσφυγες στην Ιορδανία. Αλλάζουν οι κανόνες καταγωγής ε, για την Ιορδανία για να διευκολυνθούν οι κανόνες ε, ένταξης. Η συγκήτρια. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Αυτά που είπε ο προλαλής σας. Απλώς να πω ότι η Ιορδανία είναι η πιο ευρωπαϊκή από τις χώρες του κόλπου. Και σίγουρα μπορούμε να αναλάβουμε όσο υπόθηκαν. Πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο επιστρέφεται και κυρίως ότι αποτελεί το 10% των αναγκών. Πρόκειται για ένα ποσοστό λοιπόν, αλλά όχι για το σύνολο. Βεβαίως, τα ευρωπαϊκά κριτήρια που τα συνοδεύουν με την προτεραιότητα και σίγουρα αυτά που έχουν προβλεφθεί και για άλλες χώρες πρέπει να διατηρηθούν. Σας ευχαριστώ. So, Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας θα συζητηθεί την επόμενη φορά, 6 και 7 Νοεμβρίου που θα συναντηθούμε και θα ψηφίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή και μάλλον στην Ολομέλεια θα περάσει η έκθεση το Δεκέμβριο. Έτσι ολοκληρώσαμε το σημείο 13. Στο 14 τα διάφορα υπάρχει τίποτε. Τίποτε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η επόμενη συνεδρίαση 6 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί ακριβώς και στις 7 επίσης Νοεμβρίου. Και αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση που είχα να κάνω. Καλό σας βράδυ.